Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle... Κυρίες και κύριοι, όσοι ήρθατε από εδώ, από τα μέρη μας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε ιδιαίτερα εσείς κυρία Πάρκ, αλλά και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Ιδιαίτερα βέβαια χαιρετώ τον κύριο Χόικμαρτ, γιατί είναι ο αρμόδιος για την ακρόαση εισηγητής. Καλώς ορίζω και τους προσκεκλημένους που ήρθανε να μας δώσουν συμπληρωματικές ε, πληροφορίες και ενημέρωση. Και χωρίς να βραδιπορώ, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για την ε, Επιτροπή μας αυτό του ραδιοφάσματος. Το Σεπτέμβριο είχαμε τρεις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και ε, ευρυζωνικότητα χωρίς κενά. Και αντίστοιχα τα μέτρα για, την, ε, για τα δίκτυα πρόσβασης για την προσοχή και και το πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος. Τρεις προτάσεις λοιπόν που αποτελούν τμήμα της στρατηγικής ατζέντας στα Ευρώπη 2020 και στόχο έχουμε στο θέμα αυτό να βοηθήσουμε την Ευρώπη ώστε να επεκταθεί και να αποτελέσει ένα πραγματικό, πραγματικά ουσιαστικό οικονομικό χώρο, χάρη και στο θέμα του ραδιοφάσματος. Έχουμε ήδη συζητήσει τα θέματα αυτά. Ιδιαίτερος έχουμε καταγράψει ότι υπάρχουν πολλές αποκλήσεις μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου στα κράτη-μέλη, αλλά και από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια καλύτερη κάλυψη και περισσότερη ομοιογένεια στο θέμα αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε δράση με λογικούς βέβαια στόχους για την ευρυζωνικότητα. Με την ακρόαση αυτή σκοπεύουμε να συλλέξουμε ε, πληροφορίες, ενημέρωση γιατί μέσω βράχη και μέσω πρόθεσμη προοπτική το, της χρήσης του ραδιοφάσματος. Ο κύριος Χόικμαρκ φυσικά θα, θα χωροστατήσει, αλλά φαντάζομαι και οι λοιποί συναδελφοί θα ενδιαφέρονται για τα θέματα των υπηρεσιών που μπορούν να προβλεφθούν, ε, σε ποιο βαθμό, με τι τιμήμα μπορούν να προσφερθούν αυτές οι υπηρεσίες και ποιες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ωφέλες μπορούμε να προσμένουμε από την βελτιστοποίηση του χρήσης του ραδιοφάσματος. Επίσης, θέματα ανταγωνιστικότητας και κυρίως η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εάν αρκούν τα ε, οι λωρίδες φάσματος που απελευθερώνονται, πώς μπορεί να βελτιστοποιηθεί η χρήση τους. Πολλά τα ερωτήματα όπως βλέπετε, ο χρόνος μας περιορισμένος, πρέπει όλα να λάβουν απάντηση. Και κλείνω εδώ την ε, εισήγησή μου για να μην χάνουμε άλλο χρόνο. Δίνω το λόγο στον κ. Χέκμαρτ, τον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Προέδρε, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ιδιαίτερος χαίρομαι διότι βλέπω και τους σκιώδεις εισηγητές, γιατί αρχίζουμε τώρα ουσιαστικά τη συζήτηση, αν και το θέμα έχει συζητηθεί ήδη από διάφορες πολιτικές ομάδες. Αυτή η συζήτηση για το, τη μελλοντική πολιτική για το ραδιοφάσμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί μπορεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να γίνουμε κέντρο καινοτομίας. Την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον έγινε μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Έτσι διαφημίστηκε η συνάντηση, ανάμεσα δηλαδή στην Αμερικανική και την Κινέζικη οικονομία. Το πρόβλημα με αυτή τη συνάντηση με αυτή τη σύνοδο ε, ήταν ότι βασιζόταν σε ψευδείς ε, υποθέσεις. Γιατί είναι στη δεύτερη και στην τρίτη θέση αντίστοιχα αυτές οι οικονομίες. Εμείς κατέχουμε την πρώτη θέση. we tend to uh, Ορισμένες φορές το τείνουμε να το ξεχνούμε αυτό και ή εγκαταλείπουμε τις φιλοδοξίες ε, που έχουμε. κάποιοι έχουν φιλοδοξία να ε, κατακτήσουν τη δεύτερη, την τρίτη θέση στο μέλλον. Και αυτό είναι λάθος. Εμείς πρέπει να επιδιώκουμε να είναι η καλύτερη Ευρώπη ε, και να κάνουμε αυτά που πρέπει προς όφελος της Ευρώπης. Η πολιτική του φάσματος προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία αλλαγών μεταρρυθμίσεων που μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μόνο το εξής. Ο λόγος για τον οποίο ε, χαρακτηρίζουμε την Αμερικανική και οικονομία ως τις ισχυρότερες στον κόσμο και ξεχνούμε την Ευρωπαϊκή οικονομία είναι ότι έχουν μεγάλες αγορές, μεγαλύτερες αγορές, ενώ η δική μας αγορά είναι κατακαιρματισμένη και γι' αυτό ε, τίνουμε να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε στην τρίτη θέση και αυτή στην πρώτη και στη δεύτερη. Η αγορά τηλεπικοινωνιών μας προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ε, μια ψηφιακή εσωτερική αγορά και μέσω αυτού μια πραγματική ε, εσωτερική αγορά γιατί μπορεί να ε, είναι το σημείο σε το ραδιοφάσμα. Δείτε το Google ή το Yahoo ή οποιονδήποτε άλλο φορέα. Όλες τις σύγχρονες εταιρείες ε, θεωρούμε ότι προέρχονται από τις ΗΠΑ. Οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες ποτέ δεν φαίνεται να κατακτούν το ίδιο μέγεθος, την ίδια ισχύ, γιατί δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, ε, έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα ε, στην παγκόσμια σκηνή σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, παραδείγματο χάρη. Και το ίδιο θα συμβεί με τις, ε, την κινέζικη και την ινδική βιομηχανία στο μέλλον, αν δεν κάνουμε κάτι. Πρέπει να προχωρήσουμε με τρόπο ώστε να ε, μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτή την ηγετική θέση. Και την είχαμε αυτή την ηγετική θέση για την κινητή τηλεφωνία τη δεκαετία του 90. Γιατί καταρθώσαμε να έχουμε ένα κοινό πρότυπο για τα κινητά τηλέφωνα. Μετά με σημειώθηκαν ραγδαίες εξελίξεις και από πλευράς ε, φορέων διαχειριστών των δικτύων και από πλευράς νέων συσκευών, γιατί είχαμε πολλές, ε, πολύ μεγάλη τεχνολογική πρόοδο. Δεν δημιουργείται μια νέα δηλαδή ε, αγορά τηλεπικοινωνιών, απλώς αυξήθηκε η παραγωγικότητα ε, η επιχειρηματική παραγωγικότητα και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο. Δηλαδή για τους υπολογιστές, η κοινωνία πληροφορίες, ε, η κινητή τηλεφωνία, ε, είναι τομείς που θα έχουν μεγάλη παραγωγικότητα στο μέλλον. Οπότε όταν συζητούμε την πολιτική του φάσματος, το θέμα μας δεν είναι μόνο πώς να δημιουργήσουμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την δική μας βιομηχανία ή τους δικούς μας τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Το θέμα είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, οι υπηρεσίες, οι επιχειρηματίες, όλοι εν πάση περιπτώσει στην Ευρώπη να έχουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι αυτό συνεπάγεται ευθύνε για μα. Ε, οφείλουμε να απελευθερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε το φάσμα για να έχουμε ηγετική θέση όμως, όχι για να είμαστε στην τρίτη θέση, για να είμαστε πρώτοι. Πρώτοι ως προς την καινοτομία, ως προς ε, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων νέων τομέων ε, στις ε, τηλεπικοινωνίες. Νομίζω ότι είναι μια δίρητη ανάγκη και οφείλουμε τώρα να ε, πομιστούμε την ευθύνη, γιατί αλλιώς θα χάσουμε τα πάντα. δηλαδή μπορούμε να απολέσουμε τα προνόμια που έχουμε τώρα. Δεν θα τα ξανακερδίσουμε την επόμενη δεκαετία, αν δεν κινηθούμε, και τότε θα αλλάξει τελείως το κλίμα στις τηλεπικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι τούδε γίνονται πολλές συζητήσεις για τη σύγκρουση συμφερόντων ε, ανάμεσα στην ε, τηλεοπτική ραδιοφωνική αναμετάδοση και τις νέες εμπορικές εφαρμογές ε, διαφόρων ειδών. Μα αυτό είναι λάθος. Με άλλο τρόπο θα πρέπει να συζητήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα. Πρώτον, πώς θα κατοχυρώσουμε ότι όλες οι εκπομπές πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου θα μπορέσουν να δι... χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες της ευρυζωνικής σύνδεσης. Ε, και ταυτόχρονα δεν θέλουμε να υπάρχουν φραγμοί για την παράδοση που έχουμε σε αυτές τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Μπορούμε βέβαια να αλλάξουμε τις υποδομές, αλλά οφείλουμε να μεριμνήσουμε ώστε να διατηρηθούν οι εκπομπές όπως έχουν σήμερα με ευελιξία και να έχουμε τους ίδιους στόχους, δηλαδή να απελευθερώσουμε στο μέγιστο το φάσμα, αλλά με προσοχή να ανακατανέμουμε τις ε, συχνότητες ε, και να αντισταθμίσουμε όταν χρειάζεται ε, τις απώλειες μετά την ανακατανομή του φάσματος. Και πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα και πρόεδρε... Τελειώνω σε λίγο. Αν δούμε τον όγκο των δεδομένων και πώς αυξάνεται στις τηλεπικοινωνίες, είναι αστρονομικά τα ποσά. Ε, ορισμένες φορές ε, το ξεχνάμε γιατί είναι τόσο μεγάλα και δεν ξέρουμε καν αν είναι πραγματικά ε, αυτά τα νούμερα. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια σε αυτά, αλλά ήθελα να πω ότι από τώρα μέχρι το 2014 θα αυξηθεί ο όγκος των δεδομένων θα, κατά 30, 30 φορές τουλάχιστον και στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει η μεγαλύτερη πρόσβαση για τον πληθυσμό, αυτά τα ποσά ε, ε, είναι πιο υψηλά ακόμη. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Θέλουμε να κατέχουμε την πρώτη θέση. Θέλουμε να είμαστε παρκώ ευέλικτοι, ούτω ώστε ταυτόχρονα η Ευρώπη να έχει την ηγετική θέση, αλλά και να δρομολογήσουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά για όλα τα αγαθά και τι ε, χρησιμοποιώντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την ε, διατήρηση της ε, διάδοσης του πολιτιστικού περιεχομένου μέσα από τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να κάνουμε το καλύτερο για την Ευρώπη. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε την Ευρώπη να είναι καλύτερη. Ε, μπορεί να ακούγεται αυτό προκλητικό στα αυτιά κάποιων, αλλά δεν είναι αυτό ο στόχος. Ε, όταν λέω ότι πρέπει να είναι πρώτη η Ευρώπη, δεν θέλω να προκαλέσει κάποιον. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ. Και... Έχουμε τρει πρώτου ομιλητέ, μια πρώτη ομάδα ομιλητών. Καλώ ήρθατε. Ο καθένα έχει από δέκα λεπτά και παρακαλώ να μην τα ξεπεράσετε προκειμένου να έχουμε και χρόνο για ερωτήσει. Public Policy Director της Vodafone. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί ο κύριος Παχμάχ είπε πολλά από αυτά τα οποία θα ήθελα να πω. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά τα οποία ακούστηκαν. Λέγει ο κύριος Φίζη. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το φάσμα είναι ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας σε αυτό το τμήμα της ιστορίας μας. Και μάλιστα είναι και ένας παράγοντας τον οποίο εσείς, σαν επηρεάζετε άμεσα. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες γενικότερα, τα κινητά, οι εκπομπές τηλεόρασης και όσοι χρησιμοποιούν το φάσμα, είναι υπεύθυνοι για μια τεράστια σειρά οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Και η κλίμακα, αν θέλετε, αυτών των δραστηριοτήτων και η εμβέλειά τους είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζει να αυξάνεται στο μέλλον. Ταυτόχρονα το συνολικό φάσμα το οποίο έχουμε διαθέσιμο για να στηρίξουμε αυτές τις αυξανόμενες απαιτήσεις παραμένει το ίδιο. Το μέγεθος λοιπόν του φάσματος που μπορεί να στηρίξει αυτές τις δραστηριότητες στην Ευρώπη είναι το ίδιο με αυτό το οποίο χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι. Δεν έχουμε λοιπόν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα εμείς σαν Ευρωπαίοι και δεν υπάρχει και κανένα πλεονέκτημα σε μία περιοχή του κόσμου εις βάρος μίας άλλης σχετικά με το μέγεθος του εύρος του φάσματος. Ο τρόπος είναι εμείς να βελτιστοποιήσουμε, να μέγιστοποιήσουμε τα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση της εκμετάλλευσης του φάσματος. Το θέμα είναι πόσο σωστά θα εποφεληθούμε τους συγκεκριμένους περιορισμένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και μας θέτει ακριβώς αυτό στο ίδιο επίπεδο με τους Αμερικανούς και με τους Κινέζους. Η πολιτική μας στον τομέα του φάσματος δεν ήταν θα έλεγα αυτή που θα χαρακτήριζα καλύτερη. Πολλοί θυμάστε ότι είχαμε εδώ και 10 χρόνια πληστηριασμούς 3G, οι οποίοι στην ουσία γονάτισαν σχεδόν την βιομηχανία κινητών τηλεφώνων. Αυτό άφησε εντάσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς εμπλεκομένους και σε διαφορετικά όργανα και άφησε επίσης και εντάσεις πάρα πολλές στο εσωτερικό ε, του επιχειρηματικού κόσμου. Προβλήματα τα οποία για πάρα πολύ καιρό δεν αντιμετωπίσαμε. Παρ' όλα αυτά η βιομηχανία η ευρωπαϊκή προόδευσε παρά τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε και διαχειριστήκαμε το φάσμα και όχι χάρη στον τρόπο που το κάναμε αυτό. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε την τεράστια πρόοδο την οποία έχουμε επιτελέσει, τα τεράστια βήματα προόδου τα οποία σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι συνδυασμό της RSPP, της πολιτικής δηλαδή και οι προηγούμενες ε, αλλαγές επίσης που έγιναν στο πακέτο Telecom είναι κάτι το οποίο λειτουργήσε θετικά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όμως η προσπάθεια βρίσκεται στην αρχή της ακόμα και έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Να σημειώσω δύο τομείς τους οποίους έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος και τομείς τους οποίους ε, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Οι στόχοι για το RSPP σχετικά με το φάσμα και τα ωφέλη από το ψηφιακό φάσμα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Αν θυμάμαι καλά ότι μόνο το 2008 εμείς δημοσιεύσαμε την πρώτη έκθεση σαν εταιρεία κινητών στον τομέα των κινητών τηλεφώνων που είπαμε ότι αν ξεμπλοκάρουμε αυτά τα ψηφιακά ωφέλη, τα ψηφιακά κέρδη θα έχουμε αν θέλετε 60 με 160 δις α, επιπλέον έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να γίνει η πρόταση αυτή συγκεκριμένη δράση. Πέντε χρόνια δεν είναι πάρα πολλά σε σχέση με τους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν την πολιτική μας. Παρ' όλα αυτά ήμασταν τρία-τέσσερα χρόνια πίσω από τη ΣΥΠΑ. Όταν ξεπεράσαμε λοιπόν τους αρχικούς μας φόβους και όταν ξεπεράσαμε και τις αντιθέσεις ε, που οφείλονταν στις διαφορετικές ρητορικέ των ε, κρατών μελών, μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τόσο πολύ σε αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να κληθούμε να κάνουμε στο μέλλον. Απαιτείται να κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές στην Ευρώπη, όχι μόνο στον τομέα του φάσματος, αλλά και σε άλλους τομείς, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε παγκόσμια ανταγωνιστικοί. Τα ωφέλη της αποφασιστικής δράσης είναι ξεκάθαρα. Νομίζω ότι τα κέρδη σε εισαγωγικά στη Γερμανία ε, ήταν σημαντικά πέρυσι Ήδη έχει ξεκινήσει ένα δίκτυο 4G στην Ήπεθρο χώρα με άνω των 50, με, με πολλούς σταθμούς οι οποίοι έχουν ταχύτητες, επιτρέπουν συγγνώμη ταχύτητες άνω των 50 MB ανά δευτερόλεπτο. Βέβαια στις Ηνωμένε Πολιτείες αντίστοιχες τεχνικές καλύπτουν 150 εκατομμύρια Αμερικανούς. Η Γερμανία και η Φιλανδία είναι οι πρωτοπόροι στην Ευρώπη. Όπως είπε ο κύριος Χρέχμαρκ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και ποια είναι τα ωφέλη συλλογική παρέμβαση στο σύνολο της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει να εμείνουμε στο στόχο του 2013 και ταυτόχρονα να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι όταν συζητάμε και άλλες επιλογές για το φάσμα στο μέλλον. Πρώτα θα πρέπει θα έλεγα να θεμελιώσουμε σωστά την πρόοδο την οποία έχουμε συντελέσει πριν προχωρήσουμε σε άλλα μέτρα. Ένας άλλος τομέας στον οποίο έχουμε θα έλεγα κάνει βήματα προόδου είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί ε, η βιομηχανία των κινητών και η δραστηριότητα γύρω από τα κινητά το φάσμα έτσι όπως είναι σήμερα. Πέρυσι το 2010 Χρησιμοποιήσαμε τον ρόλο τον οποίο έχουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνει το GSM για να προσφέρουμε και να διευρύνουμε ε, δυνατότητες υπηρεσιών ε, ευρέως φάσματος 3G στο 90% του ρουμανικού πληθυσμού. Μια χώρα όπου τα επίπεδα χρήσης ε, του ευρέως φάσματος ήταν αρκετά χαμηλά. Έτσι λοιπόν οι Ρουμάνοι μπορούν ε, μέσω της αναδιάταξης των ε, συχνοτήτων και για 5 μόνο ευρώ να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ευρέως φάσματος. Το ίδιο κάνουμε και στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούμε αναδιάταξη των συχνοτήτων στην Ιταλία σαν παράδειγμα για να καλύψουμε περιοχές της υπαίθρου οι οποίες στο παρελθόν δεν είχαν καμία δυνατότητα πρόσβασης σε ευρύ φάσμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ελπίζουμε να διευρύνουμε την κάλυψη 3G στο 90% του Βασιλείου το 2013 χρησιμοποιώντας τις συχνότητες GSM. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουμε σημειώσει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν δύο τομείς τώρα στους οποίους δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά το φάσμα το οποίο ελέγχει ο δημόσιος τομέας μια εποχή όπου η οικονομική πίεση είναι μεγάλη, είναι καλό να μην υπάρχουν τμήματα φάσματος τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ αυτό θα χρειαζόταν γιατί ε, θα έλεγα ελέγχονται από τον δημόσιο τομέα. Και τέλος, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην δυσδιαχειριστούμε κάποια προβλήματα όπως οι αξιολογήσεις ανταγωνισμού, οι οποίες προβλέπονται από την RSPP, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν πρέπει εμείς να καθυστερήσουμε τις αλλαγές στο ευρύ φάσμα, αλλαγές τις οποίες χρειάζεται η βιομηχανία, βιομηχανία την οποία χρειάζονται οι επενδυτές τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει οι αξιολογήσεις αυτές να γίνουν σύμφωνα με τα ίδια standards που ίσχυαν μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τώρα ξαφνικά ένα νέο διακανονιστικό πλαίσιο. Και τέλος, οι υπερβολικές τιμές για το φάσμα είτε ε, ανανεώνεται η δυνατότητα χρήσης του είτε διατίθεται για πρώτη φορά μπορεί να υπονομεύσει τα βήματα προόδου που έχουμε κάνει. Όλοι γνωρίζουμε τα οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη σήμερα. Αλλά να χρησιμοποιούν το τίμημα για τη χρήση του φάσματος για να τονώσουν την οικονομική τους ανάκαμψη είναι στρεβλό. Οποιαδήποτε λογιστικά βραχυπρόθεσμα πλεονεκτήματα στα δημοσιονομικά θα έχουν σημαντικότατο κόστος για το οικονομικό μακροπρόθεσμο μέλλον της Ευρώπης. herzlich und darf Ευχαριστώ θερμά. Και για να μην χάσουμε όλο χρόνο, παρακαλώ την κυρία Κάθριν Σπάτσια, αν δεν κάνω λάθος την προφορά του όνομα της, της να μας δώσει τις πληροφορίες. Sorry. Thank you much. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα. Δεν θα σας καταπλήξω με αυτό που λέω. Γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη ε, και συνθετική οργάνωση του BBC. Θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά και θέλουμε να υπηρετούμε τον πελάτη μας, ο οποίος απαιτεί το καλύτερο, την καλύτερη υπηρεσία. Είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Σήμερα λοιπόν επίσης θέλουμε να δραματίσουμε και το ρόλο μας για τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση. Και θέλουμε να κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες της ευρυζωνικότητας, ε, αλλά και η καλή γραμμική τηλεόραση μπορεί να κάτσει κανείς στην, ε, στο σαλόνι του και να παρακολουθήσει. Έχουμε δει πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση και αυτό που ήθελα να σας επισημάνω σήμερα είναι ε, μια μελέτη που έχουμε κάνει έτσι ώστε να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Έτσι λοιπόν. Και αυτό που θέλω να πω εγώ για το BBC και τον καταναλωτή είναι ότι ζητάει μια, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ζητάει και ευρύ ζωνικότητα και κοινή εκπομπή τα πάντα. Δεν, δεν, ε, ε, εξαρτάται μάλλον από το που βρίσκεται ο πελάτης. Ε, πίνου η αναμετάδοση, η κοινή αναμετάδοση βρίσκεται στη διάθεση του καθενό και έξω από το Λονδίνο κτλ. Εάν κανείς θέλει να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις ειδήσει, χρησιμοποιεί το smartphone του, το ευφυές τηλέφωνο. Ε, υπάρχουν οι άλλοι πελάτε οι οποίοι θα κάτσουν στι 8 η ώρα να παρακολουθήσουν τι ειδήσει στο κύριο δελτίο στην τηλεόρασή του. Οι άλλοι που θα παρακολουθήσουν τι πρόσφατε εξελίξει από το ίντερνετ. Μια ιστορική ταινία ή ένα ντοκιμαντέρ μπορεί να θέλουν να το δουν κάποια στιγμή στη βραδιά του που θα έχουν ε, το χρόνο με το σύστημα του catch-up ή με, το, ε, με τις υπηρεσίες που προσφέρει ευρυσονικότητα. Ταυτόχρονα όμως, ε, εάν βρίσκονται κάπου σε κάποιο μέρο του κόσμου που συμβαίνει κάτι σημαντικό μπορεί να θέλουν να μας στείλουν εμά στο BBC ε, κάτι ενδιαφέρον, κάποιο μικρό βίντεο και αυτό αρχίζει να ε, πολλαπλασιάζει το φαινόμενο όλο και περισσότερο. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα αλλά και τόσο αργά όσο καταναλωτής. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις εναλλακτικέ που ζητάει ο καταναλωτής. Και σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο η κύρια πλατφόρμα παραμένει η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, το κύριο μέσο, μέσον δηλαδή για το 45% των νοικοκυριών, κύριο μέσον για τηλεόραση, αλλά ταυτόχρονα και η πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιούν πολλοί από τους πολίτες μας για να λαμβάνουν σε δευτερεύους συσκευές τηλεοπτικό σήμα. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει τη μετάβαση για το 1 τέταρτο των ε, νοικοκυριών. Στο 100% θα φτάσουμε περίπου το 2012 ή το 2013. Μέχρι τώρα συμφωνώ ότι τα πράγματα πήγαν σχετικά απρόσκοπτα, απλά, ακριβώς επειδή αφήσαμε το χρόνο που χρειαζόμασταν για να προετοιμαστούμε σωστά. έχουμε προχωρήσει στην DVTB στο, και στη δεύτερη φάση προσφέροντας πολύ καλή αποτελεσματικότητα φάσματος, 65% πρόσθετη χωρητικότητα αν χρησιμοποιούμε την ε, δεύτερη γενεά και με το 50% μπορούμε να μειώσουμε την χωρητικότητα που χρειαζόμαστε για μια ε, υπηρεσία κατά 50%. Άρα κοιτάμε πλέον το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του φάσματος. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα μπορέσουμε σύντομα να απελευθερώσουμε όλο το φάσμα που χρειαζόμαστε για τις... Γιατί μπορούμε να έχουμε τις ε, καταλληλότερες λύσεις για τον κάθε καταναλωτή χάρη σε αυτό. Μπορούμε να έχουμε και εξυπηρέτηση των στόχων δημόσιας υπηρεσίας, καλύτερη παροχή υπηρεσιών ε, στοχευμένων από ότι με την ε, δορυφορική έχουμε ε, την ε, εξασφάλιση της λήψης ακόμη και για αυτούς που δεν μπορούν να έχουν ε, μια κοινή κεραία η δορυφορική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολύ καλή ανταγωνιστικότητα. Η ψηφιακή επίγεια τηλεόραση, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα, είναι μια γερή πλατφόρμα, επιτρέπει και δωρεάν υπηρεσίες και ε, επιπληρωμή, ακριβώς επειδή είναι ανοιχτή η πρόσβαση. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν τώρα να καταργηθούν σταδιακά αυτές οι υπηρεσίες της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Τώρα προχωρούμε, όπως είπα, στην μετάβαση μας και στα μισά αυτής της μετάβασης με μια, θα έλεγα, μία αποτελεσματική ε, οργάνωση μία αποτελεσματικό συντονισμό, το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρεί προς την μετάβαση αλλά με μια καθυστέρηση γιατί σκοπεύαμε το, 63 με 68 κανάλια να τα διαθέσουμε σε πληστηριασμό. Κατά τη διάρκεια όμως αυτής της διαδικασίας μας είπαν ότι πρέπει και το 61-62 να απελευθερώσουμε, πράγμα που πράξαμε. Άρα γνωρίζουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να απελευθερώσουμε μεγαλύτερο μέρος του φάσματος, ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχει και το τίμημα Στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να απελευθερώσουμε δύο κανάλια για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, ενώ έχουμε κατασκευάσει ήδη το νέο δίκτυο και το δίκτυο για τα μικρόφωνα, που σημαίνει λίγο πολύ ε, για τον καθέναν ε, στην χώρα, γιατί όλοι λίγο πολύ εξαρτώνται από τα ε, ασύρματα μικρόφωνα κάποια στιγμή και κάθε μέρα. Αυτό θα κοστίσει περίπου 120 με 122 εκατομμύρια και αν προσθέσουμε και τα μικρόφωνα ε, θα πρέπει να υπολογίσουμε άλλα 30 εκατομμύρια. Άρα, χρόνος χρειάζεται για να ρυθμιστούν αυτές οι υπηρεσίες, που είναι μεγάλο επίτευγμα. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τελειώσει μέχρι το 2013, είναι αδύνατο μάλλον για το Ηνωμένο Βασίλειο. Για το 2015 πιστεύουμε ότι είναι πιο λογική η προθεσμία για όλη την Ευρώπη. Αν λοιπόν ήταν δύσκολο το θέμα της εκαθάρισης ε, των 800 ε, μέγα, που δεν είναι ουσιαστικά η καθάριση, είναι μεταβίβαση σε άλλους χρήστες, τα 700 αυτό θα απαιτήσει πλήρη ανασχεδιασμό του, των ευρωπαϊκών δικτύων ε, επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, όχι μόνο του Βρετανικού. Ένα τεράστιο εγχείρημα, χωρίς να υπάρχει εγγύηση της ίδιας κάλυψης, δηλαδή κάποιοι περίπου το 1 τέταρτο του πληθυσμού μας, της Ευρώπης δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσουν απώλεια υπηρεσιών, επίγειων υπηρεσιών και θα χρειαστεί τουλάχιστον 50% των οικοκυριών να κάνουν κάποια αναπροσαρμογή, είτε απλώς αναζήτηση καναλιού, είτε νέα ε, κεραία και ούτω καθεξής. Άρα γενικά θα χαθεί κάποιο κομμάτι αυτής της υπηρεσίας που λέγεται τηλεόραση. Δεν λέω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απλώς θα χρειαστούμε χρόνο. Είναι ένα περίπλοκος ο σχεδιασμός η ε, ε, αναδημιουργία. Θα χρειαστεί και επικοινωνιακή πολιτική και υποστήριξη του καταναλωτή και όταν, οργανώνουμε αυτή τη διαδικασία πρέπει πάντα να εξετάζουμε τι τους αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσε αυτό ενδεχομένως να φέρει ως προς την αποτελεσματικότητα των εργασιών μας. Γιατί το πρόβλημα, εμείς το βλέπουμε ξεκάθαρα, το πρόβλημα δεν είναι να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ή μικρότερο κομμάτι, μεγαλύτερο ή μικρότερο κομμάτι του φάσματος για τις εκπομπές αλλά το να δούμε πότε, εάν, εάν μπορέσουμε ποτέ, να μετακινηθούμε προς άλλους μηχανισμούς α, υπηρεσίας και δει την ευρυζωνικότητα για τους πάντες. Ο κίνδυνος και το κόστος λοιπόν είναι σαφέστατη. Τα ωφέλη όμως, τα ωφέλη έχουν αποδειχθεί. Και με αυτό το ερωτηματικό εμείς θα θέλαμε να κάνουμε μια πραγματική μελέτη και να αντιληφθούμε τι σημαίνει, τι ανάγκες υπάρχουν ε, για νέες υπηρεσίες, τι υπηρεσίες θα, θα χρησιμοποιούμε στις επόμενες δεκαετίες, τι, θα ζητήσει, τι είδους φάσμα θα χρειαστούμε, που, ποιες ζώνες, το UHF, ζώνη πάνω από το 1 γίγα ενδεχομένως. GHz. Δεν ξέρω αν υπάρχει τουλάχιστον για τις κινητές υπηρεσίες ευρυζανικότητας ε, σαφής επιλογή. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι μας να κοιτάξουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που θα χρειαστούν οι ε, καταναλωτές στα επόμενα χρόνια, 5, 10, 20 χρόνια, ώστε να έχουμε εξασφαλίσει αρκετό φάσμα. και αρκετέ υπηρεσίε. Άρα, εάν θέλουμε μια πολιτική στηριγμένη, όπω θεωρούμε ότι είναι καλύτερο, σε γνώση ουσιαστική των δεδομένων και έρευνα της πραγματικότητα, θα πρέπει και με τις βέλτιστες πρακτικές να δουλέψουμε και με, το, με την απόδοση που μπορεί να έχει αυτή η εκαθάριση φάσματος που όπως είπα έχουμε καλές επιδόσεις από, από το 800 MHz και όπως είπαμε, ίσως να προχωρήσουμε στην καθάριση των 700 MHz στον Αμένο Βασίλειο προς το παρόν και θα θέλαμε επίσης να δούμε ε, κατά πόσον υπάρχει όφελος σε σχέση με το κόστος ε, από την εκαθάριση αυτής της, ε, αυτού του κομματιού του φάσματος. Τα ωφέλη όμως από την μετάβαση μπορεί λόγω υπερβολικά ραγδαίας εξέλιξης να ματαιωθούν. Εμείς λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε προσεκτικά με βάση τα όσα ζητάει ο καταναλωτής, ο πελάτης και με αντίτιμο, μάλλον με ε, αντιστάθμισμα ουσιαστικό. Και αυτό δεν σημαίνει οικονομικό μόνο κέρδος, αλλά και κοινωνικό και πολιτιστικό. Βεβαίω και η κινητή τηλεφωνία, η κινητή ευρυζωνικότητα και όλα αυτά έχει την δική της αξία και τη δική της προσφορά. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες ε, ευρυζωνικότητας που έχουν σημασία για τον πολίτη να εξασφαλιστούν μαζί με την διανομή, την ε, εκπομπή μάλλον μέσω επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η επιλογή περισσότερης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να σχετίζεται και να πρέπει να εξαρτάται μάλλον από στόχους δημόσιων αξιών και για την απελευθέρωση φάσματος στο μέλλον. Όπως είπαμε, πιστεύουμε ότι μπορούμε μέχρι το 2015 όλοι να έχουμε απελευθερώσει τα 800 MHz. Τουλάχιστον το 2013 για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ε, στόχος εφικτός από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε περισσότερο τώρα. Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Μεταβίβαση των 700 MHz. Αυτό μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα, αλλά είναι μακριά αυτό το βήμα. Και θα πρέπει επίση να κοιτάξουμε τι θα πρέπει να κάνουμε στο υψηλότερο μέρος του φάσματος. Αυτό είναι ένα βήμα το οποίο ήδη πρέπει να αναλυθεί. Όλα τα κομμάτια του φάσματος μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Υπάρχουν ε, κομμάτια που μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα ή που δεν χρησιμοποιούνται καθόλου ή που φερειπίν μπορούν να είναι καταλληλότερα για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συγχωρητικότητας. Άρα ας κοιτάξουμε τις πραγματικές ανάγκες, τις, ε, την καλύτερη εξέταση των ε, αναγκών αυτών, την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και το χαμηλότερο φυσικά δυνατό κόστος. Και θα ήθελα να μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για το κόστος. Το κόστος θα πρέπει αυτός που θα ωφεληθεί από την, από την εξέλιξη να το ε, επομιστεί. Τι σημαίνει αυτό. Όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορέσαμε να καθαρίσουμε τα 800 MHz με κάλυψη του συμπληρωματικού κόστους ε, από το κράτος και από τους σταθμούς. Θα πρέπει και περαιτέρω, εάν υπάρξει περισσότερη αξία από την απελευθέρωση και διάθεση σε άλλες υπηρεσίες του φάσματος, Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αυτέ οι, υπηρεσίε που χρησιμοποιούν τώρα το φάσμα απαξιώνονται τελείω. Θα πρέπει όμω να δούμε αν η αξία του είναι ικανοποιητική, αν αυτή η απελευθέρωση δηλαδή ε, προσφέρει περισσότερη αξία, εάν το κόστο νομιμοποιεί την επιπλέον επιβάρυνση και αν αυτό ισχύει τότε με ένα καλό σχεδιασμό και με ορίζοντα 20-30 ετών να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Σάιμον Φόρτ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Είναι τιμή και προνόμιο για μένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου ζητάτε. Σε 10 λεπτά πρέπει να σας πείσω ότι ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το ραδιοφάσμα τα τελευταία 125 χρόνια όταν ε, πρωτοέπαιξε ο κύριος Χέρτζ με τις ε, ραδιοσυχνότητες, έχει σημειώσει κάποια πρόοδο και ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις βασικές αξίες, να τις προσαρμόσουμε μπορούμε, να, μπορούμε και μπορούμε να διαχειριστούμε με πολύ πιο ευέλικτους τρόπους τον, ε, το ραδιοφάσμα λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων που έχουμε όλοι με τους υπολογιστές. Για να δω αν δουλεύει αυτό, δεν δουλεύει. Θα ήθελα να, να, σας, να αρχίσω με τη μελλοντική χρήση του φάσματος και να δούμε αν γίνεται ορθά η κατανομή των συχνοτήτων. Επίσης ε, θα δούμε κάποιους νέους τρόπους κοινή χρήσης του φάσματος και ε, τέλος θα μιλήσουμε για τις οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη με τις αλλαγές ε, στο ραδιοφάσμα, μιλώντας όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την κοινωνία και φυσικά για τις μικρές καθώς και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ah, this is graph which I've... Λοιπόν, αυτό, αυτή τη... αυτό το γράφημα ε, το έχω διορθώσει πάρα πολλέ φορέ γιατί είχαμε υποτιμήσει την αύξηση του αριθμού των χρηστών. Από πλευρά ε, ζήτηση υπάρχει μεγάλη πίεση στην κινητή τηλεφωνία, παραδείγματο χάρη. Η κινητή τηλεφωνία έχει φτάσει στο επίπεδο των ε, ραδιοτηλεφωνικών εκπομπών. Έχει αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε και τελικά Εντάξει, εδώ έχουμε την παγκόσμια εικόνα, αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας ό,τι συμβαίνει εκτός Ευρώπης επηρεάζει και την Ευρώπη γιατί όλα μπούμερανγκ επιστρέφουν για τα κινητά και τους υπολογιστές. Για να δούμε λίγο διεξοδικότερα τη ζήτηση φοβερή αύξηση λόγω των αλλαγών ε, στο εισόδημα, γίνεται καλύτερα η κατανομή του πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο. We Διευρύνεται το ευρυζωνικό δίκτυο, έχουμε νέους ε, χρήστες, ε, νέα σύγκληση των δεδομένων με τη φωνή για την κινητή ευρυζωνική σύνδεση. Χρειαζόμαστε περισσότερο φάσμα για τις υπηρεσίες διαδικτύου, για το μεγάλο όγκο περιεχομένου και τώρα από προσφοράς έχουμε ένα μοντέλο που είναι αυτονόητο από πολλέ πλευρές, ε, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Γιατί? Ε, δεχόμαστε πίεση από τη βιομηχανία, από την βιομηχανία των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, από το διαδίκτυο. Μας λένε θέλουμε και εμείς ένα χώρο στο φάσμα, θέλουμε να το διαχειριστείτε διαφορετικά. Οπότε ε, ας πούμε ότι έχουμε μία συσκευή, μία υπηρεσία, ε, ένα οποιοδήποτε αγαθό που θέλω να πουλήσω στους ε, πελάτες, αλλά δεν θέλω μέσω της αδειοδότησης που θα έχω λάβει να περιορίσω τους πελάτες μου στη χρήση αυτή, αυτής της συσκευής. Οπότε βλέπουμε τα στοιχεία της ίσκο στην Δυτική Ευρώπη 37 φορές έχει αυξηθεί ο όγκος από το 2009 ως το 2014 και αναμένονται άλλες ε, μεγάλες αυξήσεις στον όγκο των δεδομένων. Ε, δεχόμαστε πάρα πολύ πίεση λοιπόν για το φάσμα. Ας δούμε τι γίνεται τώρα στην Ήπεθρο. Ε, ας δούμε τι συμβαίνει στις Ήπα. Σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ε, η χρήση του φάσματος ε, είναι στη χαμηλή χρήση, με το μπλε χρώμα. Οπότε, παρότι μπορεί να έχει πουληθεί μία άδεια στον τομέα, δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο τόπο, συγκεκριμένη περιοχή εντατικά. Οπότε μπορούμε να αναρωτηθούμε μήπως γίνεται να χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο το φάσμα. Μήπως ε, είναι τεχνητό αποτέλεσμα των δημοσίων πολιτικών μας αυτή η έλλειψη φάσματος που έχουμε. Basically, Από τότε που αρχίσαμε να ρυθμίζουμε το ραδιοφάσμα πριν ε, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πολύ εντατικότερα μετά, ε, ε, τρία μοντέλα διαχείρισης είχαμε. Είχαμε τους ρυθμιστές, αυτούς που το διαχειρίζονται και θεωρούν ότι πρέπει να έχουν περισσότερο ραδιοφάσμα οι κυβερνητικέ ή οι στρατιωτικές δυνάμεις ή το άλλο μοντέλο που λέει δώστε τα όλα στους φίλου του και ξεχάστε όλα τα υπόλοιπα. Τέλο πάντων προσπαθώ να σα προκαλέσω τώρα. Θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την άξια, έχουμε τι δημοπρασίε, έχουμε τι δευτερογενεί αγορέ ή μπορεί να πούνε κάποιοι ότι αφήστε την αγορά να αυτορυθμιστεί. Ε, μπορεί έτσι να επιτύχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά εν πάση περιπτώσει Εάν ε, δείτε τα πράγματα από την πλευρά του διαχειριστή του, δικτύου κινητής τηλεφωνίας, θα διαπιστώσετε ότι αγοράζουν το φάσμα όχι μόνο για να βάλουν μέσα τις δικές τους υπηρεσίες, αλλά για να απενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών τους. Έτσι έχουν τα πράγματα στην ε, κινητή τηλεφωνία. New view. Όταν τώρα προσπαθούμε να εξετάσουμε μία νέα προσέγγιση, μία νέα άποψη, ε, βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία μπαίνει στα δύο πρώτα ε, πρότυπα. Όχι στο τρίτο πρότυπα της ευελιξίας και της κοινή χρήσης βέβαια. Αρχίζουμε να το χρησιμοποιούμε για το Bluetooth παραδείγματος χάρη, για τα σύρματα δίκτυα. Ε, οι κινητές πληρωμές έχουν βγει σχετικές ε, ανακοινώσει από τους φορείς κινητής τηλεφωνίας. Επίσης εφαρμογέ ε, ιατρικές ε, παραδείγματο χάρη για τη χρήση του φάσματος. Μπορώ να αναφέρω επίση την ηλεκτρονική τηλεδιαχείριση διαφόρων συσκευών στο σπίτι μας. Ανοίγουμε την πόρτα του γκαράζ α πούμε μακρόθεν. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ότι ένας φορέας θέλει να απελευθερώσει το δίκτυο τρίτης γενιάς 3G βάζοντας όλα τα ευρυζωνικά δεδομένα μέσα σε μία σύρματη σύνδεση. Τέλο πάντων, υπάρχουν πολλοί τεχνικοί τρόποι ε, για να το επιτύχουμε αυτό. Δηλαδή, να μοιραστούμε το φάσμα και να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Να κρύψουμε το σήμα, παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν διάφοροι ε, τρόποι για να τοποθετηθεί το σήμα σε χαμηλό επίπεδο θορύβου ε, χρειάζονται ευφυείς μαθηματικοί υπολογισμοί για να βρει κανείς ότι το σήμα είναι εκεί, το, το τηλεοπτικό σήμα μπορεί να μην καταλάβει ότι είναι εκεί ή να το βάλουμε κάπου αλλού που δεν υπάρχει παρεμβολή και, ή να χρησιμοποιήσουμε μόνο βραχία εμβέλεια ή να αποφύγουμε ε, την ε, παρεμβολή ε, τονώνοντας το σήμα των άλλων τόσο ώστε να μην συμπέσει με το δικό μας. Πολύ έξυπνοι τρόποι για να κρύψουμε το σήμα. Δείτε και τις τελευταίες μελέτες Υπάρχουν πολλά επιστημονικά ε, στοιχεία που ακολουθούν ε, την ε, προσέγγιση αυτή για να αντικαταστήσουμε την ευρυζωνικότητα με την υπολογιστική δύναμη. Περί αυτού πρόκειται. Λογισμικό, για να βρούμε τις ραδιοσυχνότητες, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και χρόνο για να σας τα πω όλα αυτά λεπτομερώς, αλλά αυτού του είδους τα πράγματα απασχολούν την πλέον προηγμένη έρευνα ε, στον τομέα αυτό και στην Ευρώπη διαβλέπουμε πελώριες ευκαιρίες σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούν να είναι δημιουργικές, να δημιουργηθεί μια νέα βιομηχανία και να είμαστε οι πρώτοι να έχουμε την πρώτη θέση για τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα η τηλεόραση αναμετάδοσης με νέα δικτυακή τεχνολογία, σας πάω πίσω στο 1994 με τη μετάβαση Νεγροπόντε, στο ψηφιακό σήμα. Ε, στην Ευρώπη λοιπόν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ευρύτερη χρήση αυτής της τηλεόρασης, ίσως τώρα να διοργανώνονται και γίνεται μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως μας είπε μόλις τώρα η Κάθριν που δείχνει με ποιο τρόπο μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές ε, οι ραδιοτηλεοπτικές αναμεταδόσεις. Να χρησιμοποιήσουμε το ευρυζωνικό δίκτυο για να φτάσουμε σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Τα, τα εγγόνια μου. Φυσικά δεν πάρεις τηλεόραση μπροστά στο Macintosh πάνε. Ή άμα είσαι στο Ηνωμένο Βασίλειο παίρνεις το iPad και βλέπεις ε, τηλεόραση. Ε, και video on demand, δηλαδή εκπομπές ε, κατά παραγγελία που τις βρίσκουν επίσης στο διαδίκτυο. Για τις μελλοντικές ε, κατευθύνσεις τώρα. Ποιοι είναι οι στόχοι. Πρώτον, πρακτικές εναλλακτικέ λύσεις. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό μας μήνυμα για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τις παρεμβολές που σας εξηγούσα να έχουμε μια κοινή συλλογική χρήση επωφελή για κάθε χρήστη. Ε, απευθύνω λοιπόν την εξή έκκληση εδώ. Εάν επιλέξουμε να έχουμε ένα μεγάλο χώρο που θα δώσουμε ε, για τις ευρυζωνικές ε, ε ασύρματες συνδέσεις, για τις δημόσιες υπηρεσίες, είναι προφανές ότι θα έχουμε χαμηλό κόστος, θα ε, και με τα 600 MHz θα έχουμε καλή πρόσβαση και στα κτίρια και θα φτάνει το σήμα σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αλλά δεν έχουμε αποφασίσει στην Ευρώπη, δεν έχουμε αποφασίσει ότι θα μοιραστούμε πολύ περισσότερο το φάσμα για να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο. Ε, δηλαδή, πολύ ενδιαφέρουσα θα ήταν η περιοχή των 600 GHz παραδείγματο χάρη. Τώρα, εντάξει, θα είμαι πάλι προκλητικό. Έχω φτιάξει ένα σενάριο που το είχαν προετοιμάσει πριν από πολύ καιρό για μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Μα ζήτησαν για εξετάσει τι μελλοντικέ εξελίξει του φάσματο. Ε, ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό που θα σας δώσω, ίσως και δεν είναι. Τι λέμε. Ότι δεν χρειάζεται άδεια για την κοινή χρήση μπορεί να αυξηθεί τα επόμενα 15 χρόνια για να καλύψει ή για να είναι διαθέσιμο σε, σε μεγαλύτερο κομμάτι του φάσματος. Αν υποκύψουμε τώρα στο μοντέλο αυτορύθμισης αγοράς δημοπρασιών και δευτερογενών ε, αγορών, ε, νομίζω ότι είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι ότι θα λειτουργήσει λέει, το σύστημα τώρα. Εάν δω τι έγινε το 2000, πάνω από 95% του φάσματος ε, το διαχειριζόμασταν από κοινού. Το 2010 έπεσε το ποσοστό σε 22%. Οι μηχανισμοί της αγοράς καλύπτουν περίπου το 72%. Κάποιοι ισχυρίζονται, έτσι. Ε, το ενδιαφέρον κομμάτι είναι αυτό που δεν χρειάζεται άδεια. Αυτό αυξήθηκε από το 4,3% στο 16,9%. το ενδιαφέρον ερώτημα είναι πρέπει να αυξηθεί πολύ περισσότερο για να πάρουμε την απόφαση ή τηλεπικοινωνίες που βλέπαμε στο προηγούμενο γράφημα, λέγαμε ότι το 30% μπορεί να είναι αντικείμενο κοινή διαχείρισης. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει επικάλυψη, δεν μου αρέσουν και οι όροι που χρησιμοποιώ, αλλά τέλος πάντων, ε, αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, επικαλύψεις θα γίνουν, δεν γίνεται κάτι άλλο. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για καινοτομίε, νέε θέσει απασχόληση. Αυτό είναι το μελλοντικό ραδιοφάσμα. Μπορούμε να αυξήσουμε το κεφάλαιό μα και αν δω ε, δημοσιεύματα σε έγκαιρα περιοδικά. Ε, ε τα μου έρχονται συνέχεια δωρεάν περιοδικά, πολύ καλά δεν λέω για τεχνικά περιοδικά. Τέλος πάντων πιστεύουν ότι δημιουργείται μια νέα τεχνολογία. Είναι δύσκολο βέβαια κάποιος να εισέλθει σε αυτή την αγορά γιατί πρέπει ταχύτατα να κατοχυρώσει τη θέση του και με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να μειώσουμε το ψηφιακό ε, χάσμα και δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στα χρηματοπιστωτικά, ε, στα, στη μηχανική, τέλος πάντων ε, θα δώσουμε το βάρος ε, στον ηλεκτρονικό ε, εξοπλισμό στους υπολογιστές και θα καλύψουμε ένα κομμάτι του ψηφιακού χάσματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική προσέγγιση η ε, παρεμβάση σα. Πολλέ πληροφορίε. Φαντάζομαι οι συναδελφοί θα έχουν ερωτήσει. σω ο κύριο Φέκμαρκ πρώτο. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να υποβάλω την ίδια ερώτηση και στους τρεις ομιλητές. Τι θα πρέπει ακριβώς να κάνουμε. Κάποια πράγματα που εσείς θα θέλατε να μην κάνουμε, ας πούμε ότι δεν τα κάνουμε. Αλλά τι άλλο θα κάνουμε στη θέση τους. Αν είναι να τα αφήσουμε όλα ελεύθερα και αν αυξηθεί γενικά η κυκλοφορία με τα κινητά με πολύ σημαντικό τρόπο. Και αν θέλουμε να καλύψουμε τη ζήτηση αυτή, τότε θα ήθελα να μου δώσετε παραδείγματα για το τι πρέπει να κάνουμε. Ο τελευταίος ομιλητής αναφέρθηκε σε μία λύση. Η λύση αυτή θα επαρκεί Η αύξηση, θυμίζω, δεν θα είναι σε τοπικό μόνο επίπεδο, αλλά θα είναι αύξηση κίνησης και ανάμεσα σε απομεμακρυσμένες περιοχές. Το παράδοξο είναι ότι όσο περισσότερη αύξηση έχουμε στις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές, τόσο αυξάνονται και τα κινητά τηλέφωνα. Είπαμε ότι όσο αυξάνεται η χρήση των σταθερών γραμμών, τόσο αυξάνεται και η χρήση των κινητών τηλεφώνων. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μετακινούμε κίνηση από τα κινητά στα σταθερά ή τούμπαλιν. Λοιπόν, πείτε μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Τροτμάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον τελευταίο ομιλητή ο οποίος αναφέρθηκε για την κατανομή του φάσματος. Εκτός αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. Εδώ πρέπει να το εμβαθύνουμε λίγο το θέμα. Νομίζω ότι για να στηρίξει κανείς την καινοτομία και για να προχωρήσει ακόμα και στις λεγόμενες γνωσιακές τεχνολογίες θα πρέπει να κάνει έρευνα, θα πρέπει να κάνει καινοτομία και αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους. Κατά συνέπεια νομίζω ότι όλοι έχουν συγκεκριμένες ευθύνες και οι εκπομπής σε εισαγωγικά και οι διαχειριστές εταιριών κινητών τηλεφώνων. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε με ενεργό τρόπο έτσι ώστε να προσανατολίσουμε σωστά και το υποενικία συμφάσμα κάτω από διαφορετικούς τρόπους αλλά και το φάσμα το οποίο είναι εκτός αδειοδότησης έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτήν την ωφέλιμη για όλους ε, ε, έκρηξη της χρήσης του φάσματος. Ναι, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι σαν βουλευτής που ασχολούμαι με τον τομέα αυτό εδώ και αρκετό καιρό η συζήτηση γύρω από το φάσμα έχει και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία μου διαφεύγουν. Αυτό είναι προφανές. Πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζει κανείς πολλά προβλήματα στο να διαμορφώσει, για να διαμορφώσει ε, κάποιες απόψεις οι οποίες να είναι τεχνικά τεκμηριωμένες και οι τεχνικές εξηγήσει οι οποίες δίδονται από πλευρά σας μπορεί να είναι ικανοποιητικέ αλλά δεν είναι απόλυτα κατανοητές. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς είναι το ποια είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Όπως είπε ένας προηγούμενος ομιλητής, τα παιδιά του δεν βλέπουν τηλεόραση σε μια ε, οθόνη τηλεοπτική. Το ίδιο συμβαίνει και σε μένα όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν τα smartphones και θα χρησιμοποιηθούν ακόμα περισσότερο τα smartphones μέχρι το 2014. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι είναι απαραίτητο να επιτραπεί και να βοηθηθεί η τεχνολογική αυτή έκρηξη και να καλυφθούν οι προσδοκίες του καταναλωτή ο οποίος θέλει να χρησιμοποιεί όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν. Νιώθω λοιπόν κάπως διστακτική όταν σας ακούω να μιλάτε και για άλλες τεχνολογικές δυνατότητες οι οποίοι υπάρχουν. Την ψηφιακή τηλεόραση σαν παράδειγμα. Μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τις εξελίξεις στην κατάσταση αυτή και επίσης τις εξελίξεις και τις τάσεις στη ζήτηση παρεχομένων υπηρεσιών. Το σωστό λοιπόν θα ήταν να προσφύγει κανείς στις δυνατότητες που θα επιτρέψουν στα προϊόντα σας να αναπτυχθούν. Και θα ήθελα να πω επίσης στους ομιλητές ότι στην παρούσα τουλάχιστον φάση και βλέποντας και το ποια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιας και το Κοινοβούλιο μας οφείλει να γνωμοδοτήσει για την πρόταση αυτή, στην πρόταση αυτή, πρέπει να δούμε αν είναι δυνατόν να κατανείμουμε το φάσμα με ελαστικό τρόπο, αλλά και να δούμε επίσης ποιες είναι οι πιο σοβαρές δυνατότητες κάλυψης των μελλοντικών αναγκών. Οι εξελίξεις τρέχουν και θα πρέπει να έχουμε αρκετό φάσμα στην διάθεσή μας για να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες αυτές που θα καλύψουν, όπως είπα, τα αιτήματα των καταναλωτών. Η ζήτηση είναι μια πραγματικότητα και σύντομα η πλειοψηφία των καταναλωτών θα θελήσει να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου. Ακούσαμε πολλά για την αποτελεσματική χρήση του φάσματος, για την κατανομή του φάσματος επίσης και ε, τα ωφέλη του φάσματος στον οικονομικό τομέα. Βλέπουμε επίσης το τι κάνουν ε, τα νέα παιδιά σήμερα, τα παιδιά μας σήμερα αλλά κανείς δεν έχει πραγματικά αναφερθεί σε θέματα συντονισμού. Στην παρούσα φάση λοιπόν απαιτείται σαν πρώτο βήμα ένας καλύτερος συντονισμός των πολιτικών των σχετικών με το ευρύ φάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ένωσης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα όμως να επιλύσουμε πρώτα δύο πρακτικά ζητήματα που με ενδιαφέρουν πάντα. Ίσως μπορεί κάποιος να μου δώσει απάντηση. Προσπαθούμε πάντοτε να σκεφτούμε τι είδους νέα ζήτηση θα υπάρξει για, αυτά τα, για αυτές τις συχνότητες. Μέχρι τώρα οι συχνότητες που έχουν απελευθερωθεί, τι ζήτηση αντιμετώπισαν. Μπορεί κανείς να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί σε ένα κράτος μέλος, υπήρξε κάποια εξέλιξη από τη μέχρι τώρα απελευθέρωση. Τι περιθώριο υπάρχει. Και επίσης δεύτερη ερώτηση που σχετίζεται και με όσα είπε η κυρία από το BBC για το κόστος που προκύπτει. Προκύπτει λοιπόν κάποιο κόστος. Αυτό το ζήτημα το, της δαπάνης, εάν επιληθεί, διευκολύνει και την απάντηση που θα δώσει το BBC. Ποιος θα, ποιος θα μάλλον το κόστος, τι είδους μοντέλα προβλέπονται Ας ξεκινήσουμε και με τους τρεις, ε, με τον κύριο Φόρς καταρχάς, να ακούσουμε όμως και τους τρεις ομιλητές. Τεχνικά τα ζητήματα είναι. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα, το ερώτημα μάλλον είναι τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο μέτωπο των συχνοτήτων. Εξ όσων διαπιστώνω εγώ, και μάλλον ήδη συμβαίνει στην πράξη, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο. Οι αρχές δείχνουν ενδιαφέρον και θέλουν να προχωρήσουν περαιτέρω. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μία ομάδα εργασίας η οποία λέει ότι αν πρόκειται να ανατραπεί, όχι βράχη αλλά μακροπρόθεσμα, η ισχύουσα κατανομή φάσματος που ξέρω ότι θα προκαλέσει αγανακτισμένες αντιδράσεις ε, και τρόμο, αποτροπιασμό σε όλα τα μέλη εδώ της ομάδας, αλλά τέλος πάντων εγώ αποτολμώ το, την πρόταση. Τι θα κάνουμε? Θα κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι επιλογές υπάρχουν. Υπήρχε. Το 2007 μια μελέτη που είχαμε κάνει για την Deutsche Telekom ε, εξέτασε το ψηφιακό γεωγραφικό μέρισμα ε, με ορίζοντα το 2020. Βέβαια η μελέτα το 2007, επομένως είναι κάπως παροχημένη πια. Ε, αυτό που θα συστήναμε λοιπόν είναι τέτοιες εξελίξεις να εξετάζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα ώστε στην Ευρώπη να έχουμε την ευκαιρία να ανακτήσουμε τουλάχιστον μερίδιο της τεχνολογικής πρωτοπορίας που είχαμε στο παρελθόν στις επικοινωνίες, ραδιοτηλεπικοινωνίες ε, και τους υπολογιστές στη χρήση δηλαδή, των νέων τεχνολογιών. Άρα χρειαζόμαστε ένα φύλλο πορείας ε, που θα δείχνει πώς προχωρούμε στη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Βέβαια δεν είναι καινούρια τεχνολογία, υπάρχει γιατί δεν σας είναι γνωστή ενδεχομένω, αλλά ε, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ήδη στις, ε, σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, ειδικά οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πρωτοπόρες πάντα έχουν αξιοποιήσει και χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία. Πλην όμως αυτό που κάθεται τώρα σαφές είναι ότι αυτή η τεχνολογία θα είναι πιο διαθέσιμη στο μέλλον και άρα και με χαρά ακούω τα ερωτήματά σας. Και άρα, εάν πρόκειται να προχωρήσουμε θα πρέπει να δούμε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις πιο σοβαρά, να τις διαχειριστούμε πιο σωστά, λαμβανομένων υπόψη και των ε, συσχετισμών κόστους και ωφέλους που ανέφερε και η Κατρίνα. Και όταν λέτε ποιο πληρώνει την ύφη, ε, μα ακριβώ περί αυτού πρόκειται. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση που κάνουμε πριν από τέσσερα χρόνια πια. και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το φάσμα στην Ευρώπη. Κάνουμε λοιπόν μια ανάλυση που να κοιτάει και κυρίως στις κοινωνικές πτυχές και τις οικονομικές πτυχές και τις τεχνολογικές πτυχές και εξετάζει το, τα πλεονεκτήματα. Δουλειές, πνευματικό κεφάλαιο στην Ευρώπη ως κέρδος. Και όλα αυτά τα σταθμίζουμε και λέμε να κάπως έτσι πρέπει να προαγάγουμε το φάσμα στην Ευρώπη. Παραλίγο δεν θα τυράξουμε όλο στον αέρα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν. και να πούμε ότι έτσι θα γίνεται από εδώ και μπρος η εκπομπή στην Ευρώπη, ένα τάδε ποσοστό, αλλά ίσως και πιο χαμηλό, θα πηγαίνει μόνο στην επίγεια τηλεόραση και μετά θα υπάρχει ευρυζωνικότητα, αλλά θα χρησιμοποιείται και η ε, νέα τεχνολογία, έστω και αν δεν είναι πολύ γνωστή. Αυτές είναι διάφορες ε, επιλογέ που έχουμε τώρα, γιατί έχουμε τεράστια δυνατότητα επεξεργασία δεδομένων, αλλά χαμηλό σχετικά κόστο. Αν δούμε τα, κινικά, τα κινητά μα τηλέφωνα στο 95% έχουν μέσα ένα μικροτσίπ ευρωπαϊκό από μια μικρή εταιρεία σχεδιασμού του Cambridge. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκ τούτου, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρόκειται όμως για μια μοναδική υπογραμμίζω ευκαιρία να πιάσουμε το ε, σειρμό, να ανέβουμε στο τρένο των εξελίξεων. και ως εκ τούτου στην ερώτηση για τον οδικό χάρτη, ναι, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πολύ σαφή δεδομένα. Γι' αυτό μίλησα για τα 600 MHz και όχι τα 2,4 GHz που έχουν πολύ μεγαλύτερη δίσδυση ε, Γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες είναι προκλητική μια τέτοια τοποθέτηση. Υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητε και δυνατότητες και με κάποιο τρόπο πρέπει να τις συγκεράσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σμάτσα. Λοιπόν, για τις υπηρεσίες που με ρωτήσατε. Μιλήσατε Μίλησαν όλοι μάλλον για τους ε, νέους ε, που διαβάζουν ό,τι βρουν στο ίντερνετ χρησιμοποιώντας ε, τους κινητούς υπολογιστές τους. Όταν τους αρέσει όμως μία εκπομπή θέλουν να το δουν στην οθόνη υψηλής ευκρίνειας και σε τρεις διαστάσεις 3D αν γίνεται για τις υπηρεσίες. Ε, το θέμα είναι πώς μπορούμε από κοινού να ε, διαχειριστούμε το φάσμα και να χωρέσουν όλες οι υπηρεσίες. Μας μιλήσατε για την ικανότητα που έχουν αυτές οι ευφυείς ε, συσκευές να κάνουν μια πιο ευέλικτη χρήση του φάσματος και αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το ερευνητικό τμήμα μας στο BBC μελετούν αυτή τη δυνατότητα. Ακόμη δεν έχουν καταλήξει. Αν θέλουμε τώρα οι συσκευές αυτές να χρησιμοποιούν το φάσμα και να υπάρχουν επικαλύψεις με άλλους χρήστες χωρίς όμως να έχουμε παρεμβολές, δεν χρειάζεται πολύ έρευνα. Όμως θα θα χρειαστούν ισχυρά πρότυπα, τεχνικά πρότυπα, γιατί αλλιώς θα γίνει ένα μπάχαλο και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τίποτα από το φάσμα. Λοιπόν, δεν θέλουμε να, από την παραδοσιακή αυτή προσέγγιση, αποφασίσω και διατάζω να περάσουμε στην φιλελεύθερη προσέγγιση απευθείας, ε, χωρίς καμία ρύθμιση. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι με τις ε, δημοπρασίες θα βγάλουμε μακρύ. Με τους πληστηριασμούς αυτούς ε, στις 27 χώρες ε, δεν έχουμε καλές πιθανότητες να πετύχουμε. Χρειάζεται εναρμόνιση, χρειάζεται συντονισμός για να έχουμε καλή χρήση του ραδιοφάσματος. Έχουμε ελάχιστες πιθανότητες λοιπόν με την παλιά προσέγγιση. Αν χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση της συλλογική χρήσης, common approach, τότε θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την σωστή χρήση του φάσματος. Βέβαια, ίσως δεν λειτουργούν ακριβώς όπως πρέπει τώρα οι συσκευές, αλλά αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε εναρμόνιση και χρειαζόμαστε κοινά τεχνικά πρότυπα. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Βέβαια, μπορεί να διατηρήσουμε εν μέρει την προσέγγιση μας, τον έλεγχο, έτσι, να ελέγχουμε το φάσμα για να έχουμε τη βέλτιστη αξία. Να χρησιμοποιήσουμε όλο τον ειδών της ευθύς ε, συσκευέ, ε, να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Ε, χρειαζόμαστε τις κινητές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα όμως χρειαζόμαστε ισχυρές σταθερές γραμμές για να έχουμε την τηλεόραση σε, τρίτη, σε τρεις διαστάσεις, να το βλέπετε το μάτι σε τρει διαστάσει. Αυτό δεν γίνεται μέσα από το ευρωζωνικό δίκτυο. Σίγουρα μπορώ να σας το πω, σχεδόν σίγουρα μπορώ να το ισχυριστώ. My, my uh, κύριος Φίζη. Ε, εύκολο είναι να πάει κανεί στις γραφικές παραστάσεις, στις γνωστές γραφικές παραστάσεις της ΣΥΣΚΟ και να πανικοβληθεί και να πει όχι θα πάθουμε κρίση φάσματος». Δεν έχουμε αρκετή χωρητικότητα για να εξυπηρετήσουμε όλη τη ζήτηση. Και αυτό θα ήταν αλήθεια αν δεν είχαμε κάνει κάτι τα τελευταία τρία με πέντε χρόνια σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στην πολιτική για το φάσμα. Εδώ και πέντε χρόνια βρισκόμασταν σε μια εξαιρετικά κακή κατάσταση σχετικά με το φάσμα, αλλά δεν θα πρέπει να πανικοβαλόμεθα. Δεν υπάρχει μια πραγματική κρίση εφόσον εφαρμόσουμε και εκτελέσουμε σωστά τα βήματα και τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να δημιουργούμε. Υπάρχει αρκετό ε, φάσμα για την βιομηχανία των κινητών το οποίο είναι υποεκμετάλλευση και η πρόκληση είναι να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή των αποφάσεων τις οποίες έχουμε ήδη πάρει. Ανησυχώ ιδιαίτερα όταν λέμε ότι από το 2013 μπορούμε να γλιστρήσουμε το στο 2015, γιατί τα επόμενα τρία χρόνια είναι μια κρίσιμη περίοδος. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα όμως σαν βιομηχανία για τη βελτίωση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε και σε επίπεδο υποδομών στα κτίρια και σε σχέση με τον τρόπο που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες. Έχουμε ακούσει κάποιες πληροφορίες από πλευρά στη ΣΥΣΚΟ, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία μας δίνουν την δυνατότητα να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και μάλιστα με τον τρόπο αυτό λειτουργούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εφόσον λοιπόν συνεχίζουμε με την ίδια θα έλεγα τακτική δεν απειλούμεθα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε είναι σε 27 χώρες ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης αν θέλετε και εφαρμογή των μέτρων τα οποία έχουμε αποφασίσει. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Πρέπει λοιπόν η εκτέλεση των συγκεκριμένων μέτρων και αποφάσεων να γίνεται έγκαιρα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πράγματι, εμείς αποφασίσαμε στην Ευρώπη, ξεχάστε λίγο τα 700 MHz και τα λοιπά. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν έλεγα στην Ευρώπη μετά από μια καλή συζήτηση που κράτησε και πολύ καιρό στο ότι θα πρέπει εμείς να διαθέσουμε ε, και σε άλλα επίπεδα φάσματος κάποιες δυνατότητες στον ιδιωτικό τομέα και παρόλα αυτά Μόνο σε μία μόνο μεγάλη χώρα σήμερα έχει γίνει κάτι τέτοιο. Απαιτείται λοιπόν σε όλες τις άλλες χώρες, με την εξαίρεση όπως είπα της Γερμανίας και της Φιλανδίας, να συνεχίσουμε με την εφαρμογή των αποφάσεων τις οποίες έχουμε συζητήσει επί τρία ολόκληρα χρόνια. Κατανοώ βέβαια το ενδιαφέρον της Κάθρινς για το θέμα ότι θα πρέπει δηλαδή να έχουμε τα επόμενα χρόνια συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα είναι και τι μορφή θα έχει το επόμενο ασπέκτρουμα. Αλλά όμως τα, τελευταία, τα επόμενα λίγα χρόνια έχουμε την δυνατότητα να βελτιώσουμε τα πράγματα επί τη βάση όσων έχουμε αποφασίσει και αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει πρέπει να γίνουν πραγματικότητα και πρέπει να γίνουν πραγματικότητα σε μια υγιή οικονομική βάση και κυρίως έγκαιρα. Δεν θα πρέπει το κόστος για τις επιχειρήσεις να είναι τόσο υψηλό όσο ονειρεύονται ε, μερικές φορές οι ε, κυβερνήσεις. Λοιπόν, το πόσες από τις αποφάσεις τις οποίες έχουμε λάβει μέχρι τώρα έχουν ήδη εφαρμοστεί είναι το ερώτημα το οποίο ε, τίθεται και θα τίθεται για τα επόμενα χρόνια. Όταν δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε για το επόμενο φάσμα. Τι συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι αλλαγές έγιναν επί τη βάση του ότι εμείς που εκπέμπουμε δεν θα έπρεπε να απελευθερώσουμε τα 800 MHz. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί η κυβέρνηση και η ΟΦΚΟ η ανεξάρτητη αρχή, πήρε αποφάσεις χωρίς να διαβουλευτεί ουσιαστικά. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το φάσμα όταν χρειαστεί, αλλά παρόλα αυτά καλό θα ήταν να μπορέσουμε να το κάνουμε ε, όταν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα τα οποία μας ζητήθηκαν από πλευράς ε, του ρυθμιστή και της κυβέρνησης. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν ότι απαιτείται να εφαρμοστούν σε μία πρώτη φάση με σωστό τρόπο και έγκαιρα οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Και τις απαντήσεις σας, την ενημέρωση που μας δώσατε. Κλείνουμε έτσι τον πρώτο γύρο ομιλητών. Ευχαριστούμε τους προσκεκλισμένους μας και παρακαλώ τους επόμενους ε, ομιλητές. Και βέβαια αναλαμβάνει και ο Γκέναρτ την ε, καθοδήγηση των συνομιλιών. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. So, may I ask the new panel to take their seats. Παρακαλώ τώρα τους προσεχείς απολυτές να καθίσουν στις θέσεις τους. As we met earlier. Hello. Yes. Nice to see you again. And uh, Denise Leskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, here. He's here. Hello. So, thank you very much, and I think we will um, start this part of the hearing. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε αμέσως το δεύτερο αυτό κομμάτι της ε, συζήτησης με ένα θέμα το οποίο ακούσαμε ακροθυγός από, τους, ε, από την πρώτη ομάδα μιλητών. Ίσως μπορούμε να βαθύνουμε περισσότερο η συζήτηση είχε να κάνει με το πώς βλέπουμε την κατάσταση για το μέλλον. Δηλαδή δυναμικό ή δυνατότητε για το μέλλον. Ο κύριο Κρίστοφερ Γκάου, τώρα επικεφαλή τη πολιτική για το φάσμα τη ΣΥΣΚΟ, παρακαλώ. Δέκα λεπτά ο καθένα. Και θα καταλάβετε από την έκφραση στο πρόσωπό μου ότι εξαντλήσατε το χρόνο σας. So, um, Στόχος αυτού του πάνελ είναι να εξετάσει ακριβώς τις μελλοντικές δυνατότητες για το φάσμα στο μέλλον και πώς επηρεάζονται οι πολιτικές που θα καθορίσουν το φάσμα. Θα σας δώσω κάποιους πίνακες, τους οποίους έχετε δει για αρκετές φορές θα έλεγα σήμερα, έτσι και αλλιώ η εταιρεία μου δημιουργεί αυτά τα γραφήματα που δείχνει ακριβώς το πού πηγαίνει η κίνηση των κινητών τηλεφώνων τα επόμενα χρόνια. Είναι ο πιο ενδιαφέρον τομέας τον οποίο έχουμε μπροστά μας, ο τομέας των κινητών. Αυτό που βλέπουμε ότι διπλασιάζεται κάθε χρόνο από το 9 μέχρι το 2014. Τα νέα στατιστικά για τη μελέτη αυτή θα κυκλοφορήσουν σήμερα. Συγγνώμη δεν μπορώ να σας τα δείξω από τώρα, αλλά επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή την τάση και δείχνουν ότι το 2014 δεν θα μιλάμε για 3,6 τελεμπάιτ τον μήνα, αλλά για πάνω των 5. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλότερη από αυτούς που περιμένουμε. Τι γίνεται, τι, σε τι οφείλεται αυτό στο βίντεο, βίντεο στο κινητό, βίντεο στο λάπτοπ. Λοιπόν, έχουμε τα smartphones από τη μία και τα laptops από την άλλη. Αυτό εξηγεί τη διαφορά. Αν πάρετε τα iPhone σαν παράδειγμα, δημιουργεί 30 φορές περισσότερη κίνηση από ότι ένα κανονικό τηλέφωνο. Ένα λάπτοπ 100 φορές περισσότερη κίνηση στο φάσμα από ότι ένα κινητό απλό τηλέφωνο και το ίδιο και με τα iPads ε, τα οποία θα, θα, τονώσουν αυτό, αυτή την τάση γιατί δεν τα είχαμε λάβει υπόψη τα τελευταία χρόνια βέβαια. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη και, στην ε, και στον υπόλοιπο επίσης κόσμο. Αν δείτε ε, από το κάτω μέρος θα δείτε την Δυτική Ευρώπη βλέπετε ότι το 34% του συνόλου του φάσματος θα χρησιμοποιείται στην Ευρώπη το 2014. Η Ευρώπη θα είναι η μεγαλύτερη αγορά και αυτό δείχνει ότι η Ευρώπη είναι και η μεγαλύτερη οικονομία και όχι μόνο στην διακίνηση στο φάσμα. Οι καλύτερες και ψηλότερες ταχύτητες είναι επίσης στη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε 600 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, ε, ε, κιλομπίτ, συγγνώμη, αναδευτερόλεπτο στην Ευρώπη και αυτό κάτι λέει σχετικά με τις πολιτικές κατανομής του φάσματος. Γιατί για να παραμείνουμε στην πρωτοπορία με υψηλές ταχύτητες πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φύση και οι, ρυθμιστές, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν συγκεκριμένο ρόλο εδώ να παίξουν. Ένας από τους ξεκάθαρους τομείς είναι ακριβώς οι αδειοδοτήσεις για ε, το ευρύ φάσμα για τα κινητά τηλέφωνα. Τα στοιχεία δείχνουν ποιες είναι οι προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται για τη διάθεση του φάσματος από την ε, πολιτική, από τα μέτρα της Επιτροπής. Προβλέπονται ε, ακριβώς τα 1800 MHz, φωνητική κινητή τηλεφωνία, Έχουμε επίσης και το σπέκτρουμ το φάσμα σε 2,6 GHz και τα λοιπά. Έχουμε επίσης και το 2,1 GHz, αλλά πάνω σε αυτό δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση και δεν προβλέπεται κάτι στα πλαίσια της RSPP. Άλλοι ομιλητές συγκέντρωσαν την προσοχή τους στο αδειοδοτημένο φάσμα. Εγώ θα σας μιλήσω για έναν άλλο τομέα. Αναφέρθηκαν και σε αυτό, ιδιαίτερο εκπρόσωπος της Vodafone βέβαια. Υπάρχουν και άλλοι χρήστες οι οποίοι ε, θέλουν να αναφερθούν σε ένα δεύτερο, ε, ε, θα έλεγα, ψηφιακό μέρισμα, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Είναι τα συστήματα πρόσβασης στην ασήμαντη τηλεφωνία και το πιο γνωστό από αυτά είναι το Wi-Fi. Εδώ ε, η, προβολή που κάνω είναι περισσότερο τεχνική θα έλεγα. Αριστερά βλέπετε το πού βρισκόμαστε σε επίπεδο των standards για το Wi-Fi και από την άλλη βλέπετε τα αναμενόμενα. Καταρχάς αυτό που λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το θέμα της ταχύτητας. Έτσι με αυτά τα πρότυπα θα έχουμε πολύ υψηλότερη ταχύτητα, 3,2 Gbps δηλαδή το δευτερόλεπτο και το δεύτερο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι το κομμάτι του φάσματος που μπορεί να απαιτείται. Από τα κανάλια 14 GHz ε, φτάνουμε στα 16 MHz ε, και επίσης το χρονοδιάγραμμα. Το πρότυπο θα είναι έτοιμο το 2013. Οπότε, αν αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε από ρυθμιστική σκοπιά, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και το πρόγραμμα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πάρα πολύ καλό εφαλτήριο. Προς το παρόν. Όπω έχει τώρα δηλαδή το πρόγραμμα του φάσματος της Ένωσης. Γιατί ασχολούμαστε με αυτά, τι, τι χρειαζόμαστε ε, την, την υψηλότερη ταχύτητα στα ασύρματα δίκτυα, γιατί συζητούμε τα νέα πρότυπα. Υπάρχει το offloading, το επωνομαζόμενο, ε, μιλώντας για τη μεταφορά των δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία και έχουμε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία όπω σα τα έδειξα και εγώ και όπω είπε και ο κύριο Φόρτζε, ε, ε, δηλαδή ξεφορτώνεται ο όγκος των δεδομένων ε, της κινητής τηλεφωνίας στα ασύρματα δίκτυα ε, και τις περισσότερες φορές έχουμε κάποια, ε, σταθε... είμαστε σταθερό σημείο, δηλαδή είμαστε, ξέρω εγώ, είτε στη δουλειά μας είτε στο σπίτι, το 60% του χρόνου μας. Οπότε, δεν χρειαζόμαστε την κινητή τηλεφωνία συνέχεια. Θα χρησιμοποιήσω το προηγούμενο παράδειγμα για τη Mobistar. Έτσι, αν έχετε το iPhone σας, ε, παραδείγματο χάρη, χρησιμοποιείτε το δίκτυο Mobistar, αυτόματα ε, ε, εντοπίζει αν υπάρχει ένα ασύρματο δίκτυο και αυτόματα σας περνάει στο ασύρματο δίκτυο. Γιατί, διότι θέλουν η κυκλοφορία όγκου των δεδομένων στο μέτρο του δυνατού να περνάει μέσα από το ασύρματο δίκτυο, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα ε, που θα αποδοθεί στα κινητά δίκτυα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το φαινόμενο που παρατηρούν. Μπορώ να σας δώσω και ένα άλλο ε, παράδειγμα των κοινωνικών εφαρμογών. Γιατί δηλαδή θέλουμε ε, να έχουμε αυτά τα ασύρματα τα ε, δίκτυα γιατί θέλουμε να περνάνε όλο ένα και περισσότερο τα δεδομένα οπτικοακουστικά και άλλα μέσα από αυτά τα σύρματα δίκτυα. Λοιπόν, ας δούμε τα νοσοκομεία. Ένα λεπτό και θα σας βάλω όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα στην οθόνη σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλή ευκρίνεια βίντεο για να βελτιώσετε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτοματοποίηση δηλαδή, μπορούν να κατευθείαν στα τηλέφωνα των ιατρών να περνάνε τα δεδομένα. Επίσης, μπορούν ειδοποιήσεις να στέλνονται αυτόματα ηλεκτρονικά και από πλευρά ε, των βίντεο μπορούμε να έχουμε καλύτερες ε, βίντεο επικοινωνίε ε, για τους περιθάλποντες. Χρειαζόμαστε αυτές τις τεχνολογικές πρόοδους, ώστε να παρέχεται καλύτερη περίθαλψη. Λοιπόν, για την παιδεία, ένα άλλο παράδειγμα, εδώ χρησιμοποιούνται λένε και περισσότερο τα σύρματα δίκτυα μέσα στην τάξη και συνεπάγεται αυτό μεγάλο ωφέλη. Τι μπορείτε να κάνετε, να έχετε έναν πολύ καλό καθηγητή, δάσκαλο και να κάνετε μια διαδραστική συζήτηση μαζί τους από διάφορες τάξεις ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας υψηλής σε βιντεοδιάσκεψη αμφωτέρων των πλευρών. Ε, τηλεπαρουσία έτσι ονομάζεται αυτό, telepresence. Να ένα παράδειγμα από τον τομέα της παιδείας ε, και υπάρχει και το θέμα ε, της δημιουργίας οικιακών δικτύων. Στο ίδιο σας το σπίτι δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες για να παράξετε περιεχόμενο, για να χρησιμοποιήσετε ένα κλειστό σύστημα ασφαλείας ε, και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για περιεχόμενο 3D διαστάσεων, χρησιμοποιώντας βέβαια το ασύρματο δίκτυο, αλλά και στρέφομαι στην κυρία από το BBC, σίγουρα δεν θα συμβεί αυτό ε, αύριο. Χρειάζεται κάποια έρευνα για να προσαρμοστούν οι συσκευέ. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Ο κύριος Φόρτζ μας είπε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 600 MHz, ε, το μη αδειοδοτημένο ε, κομμάτι του φάσματος. Εμείς προτιμούμε τα 5 GHz, διότι είναι πιο εύχριστη, πιο άμεση λύση και δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Ε, δηλαδή στα 2,4 MHz λειτουργούν ήδη τα ασύρματα δίκτυα και στα 5 GHz. Και εμεί τι θέλουμε, αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δείτε αυτό το γράφημα, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα, τέλο πάντων κάτω αριστερά. Η Ιαπωνία, η ΙΠΑ, η Δυτική Ευρώπη και η Ινδία σε ένα ορισμένο βαθμό ήδη έχουν φάσμα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τα ασύρματα δίκτυα στα 5 GHz. Δηλαδή αυτό ήδη συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Θέλουμε να το επεκτείνουμε. Αντί να έχουμε αυτά τα δύο μεγάλα κομμάτια, ε, στο γράφημα οι πράσινε οι θέλουμε λοιπόν να διαδοθεί αυτό σε ολόκληρο το φάσμα. Ε, μέχρι τα 525 δηλαδή γίγκαχες να καλύψουμε όλη την ψαλίδα, ούτω ώστε να υπάρξει κοινή χρήση με τους υφιστάμενου χρήστες, να δοθούν κοινέ απαντήσεις στα προβλήματα και χρησιμοποιώντα ε, τεχνικέ προσαρμογής δεν θα ενοχληθούν ε, οι χρήστε, κυρίω ε, τα ραντάρ δηλαδή, οι στρατιωτικοί χρήστε και να μην παρεμποδιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δορυφόρων. θα επαναλάβω και πάλι για να θυμάστε αυτά που είπα. Ε, αυξάνεται η κινητή τηλεφωνία με ραγδαίους ρυθμούς ε, και πρέπει κάπως να ανταπεξέλθουμε ε, και γιατί ζητάμε επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου είτε μιλάμε για σύρματη πρόσβαση, για σύνδεση με σταθερό δίκτυο είτε όχι, στους τομείς ε, της υγείας, ε, της παιδείας και της οικιακής χρήση, υπάρχουν ε, πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και ε, μπορούμε να ασχοληθούμε με το αδειοδοτημένο κομμάτι του φάσματο. Αυτό είναι το αντικείμενο του προγράμματο ε, ραδιοφάσματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να ασχοληθούμε και με το μη αδειοδοτημένο κομμάτι. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ζητήσει την κατανομή 5 GHz για τα ασύρματα δίκτυα να καλύπτουν τουλάχιστον ολόκληρο το φάσμα ε, να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα, παραδείγματος Θα μπορούσατε να το ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε και θα περάσουμε ευθύ αμέσω στην ε, παρουσίαση του κυρίου Πάτρικ Φανίφτρικ για τις εφαρμογές ε, του φάσματος. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τη δυνατότητα που δίνετε να σας μιλήσω σήμερα στο πλαίσιο αυτή τη συνεδριάσεως. Μιλούμε λίγο για, την... για τις για το μέλλον και κυρίως τη ρόλο μπορούν να δραματίσουν ε, οι δορυφόροι, οι ήδη δραματίζουν. Καταρχάς λοιπόν ε, κάποια στοιχεία για το ποιοι είμαστε. Η SES, e ε, Παγκόσμιος Πάροχος Υπηρεσιών Δορυφόρου. Καλύπτουμε σχεδόν ολόκληρη την Ιφίλιο. Έχουμε την Άστρα και την Spotcast κυρίως. Η SES e δρεύει στο Λουξεμβούργο δύο ώρες περίπου μακριά από τι Βρυξέλλε. Έχουμε επίση στο Ηνωμένο Βασίλειο τη κάτω χώρες και άλλε περιοχέ τη Ευρώπη. Προσφέρουμε σε τελικό ε, δορυφορικό λοιπόν δυναμικό, βίντεο, δεδομένα, ευρυζωνικότητα, τηλεφωνία και κυβερνητικές ε, και κρατικές μάλλον υπηρεσίες, και μέσω του δικτύου Άστρα, όπως θα γνωρίζετε ίσως, ε, αγγίζουμε περίπου 150 εκατομμύρια νοικοκυριά. Έχουμε 17 περίπου, έχουμε 17 δορυφόρους που συνδέονται με τα συστήματα C, Q και K και έχουμε περιφερειακή εστίαση την Ευρώπη, παρότι είμαστε παγκόσμιο παράγοντα όπω έχουμε δραστηριότητα σε ολόκληρη την Φίλιο, αλλά να αναπτύσσουμε, όπω είπαμε, και στον υπόλοιπο κόσμο τι δραστηριότητέ μα, ιδιαίτερα στην Αφρική. Ξέρω ότι δεν είναι ευανάγνωστες αυτές οι διαφάνειες για όλους όσοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε κυρίως την παρουσία των ε, δορυφορικών υπηρεσιών, κατά 75 περίπου ε, δορυφορική πλοήγηση και ούτω καθεξής ε, δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, δηλαδή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων μας, 75% περίπου. και 115 εκατομμύρια. Ο δορυφόρο λοιπόν, δυνατότητε για το μέλλον. Ο δορυφόρο μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερε δυνατότητε για το μέλλον. Έχει πάρα πολλέ δυνατότητε σε εφαρμογέ με δύο τρόπου. Είτε με, τις, ε, με την παροχή ακριβώ αυτού του δυναμικού τη ικανότητα μπορεί να υποδεχθεί μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις και για τον καταναλωτή ε, τη διανομή της κοινή ε, τηλεόρασης αλλά και της επίγειας ψηφιακής, προσθέμενη αξία και ευρυζωνικότητα. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω εδώ. Ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε στις υπηρεσίες της Άστρα για την ευρυζωνικότητα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο και είναι πιστεύω ενδιαφέρον η αποτελεσματική χρήση του φάσματος. Οι ε, δορυφόροι χρησιμοποιούν κατά πολύ αποτελεσματικό τρόπο τον, ε, το φάσμα, το διαθέσιμο φάσμα. Σας δείχνω εδώ έναν ε, δορυφόρο με κάλυψη την Ευρώπη, μία μόνο ακτίνα, ακτίδα μάλλον, που καλύπτει όλη την Ευρώπη. Μπορεί να την ξαναχρησιμοποιήσει όμως και να πιάσει Δυτική Αφρική και άλλη μια φορά και να χρησιμοποιήσει την, να, να πιάσει την Ανατολική Αφρική και με την ε, διπλή πόλωση μπορεί να διπλασιάσει, να υπερδιπλασιάσει μάλλον το φάσμα που χρησιμοποιεί. Την αποτελεσματικότητα του φάσματος που χρησιμοποιεί. Έχουμε να κάνουμε με μια χρήση η οποία και μαζί με την κινητή τηλεφωνία μπορεί να πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητά της ε, συνέχεια. Και αυτό με ε, πολλαπλασιαστικό με δυνατότητα πολλαπλασιασμού των, ε, των μεγεθών, διότι με απόκληση μίας μοίρας μόνο μπορούμε, ή και μερικών κατοστών της μοίρας μόνο, μπορούμε να έχουμε άλλο δορυφόρο και άλλη κάλυψη. άρα μπορούμε να έχουμε πληρέστατη κάλυψη. Και εδώ θα ήθελα να φερθώ λίγο στην ευρυζωνικότητα των ε, δορυφορών. Θα πρέπει εγώ να σας διαβάσω βέβαια τη διαφάνεια, γιατί δεν μπορείτε να διαβάσετε φαντάζομαι την αίθουσα. Λοιπόν, ε, μπορεί να προσφέρει μια άμεση λύση ως προς το ψηφιακό μέρισμα ε, ο δορυφόρος. Μπορεί να προσεγγίσει κάθε νοικοκυριό στην Ευρώπη, είτε στο αστικό κέντρο, είτε στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της Πέθρου χωρίς περιορισμό. Ήδη υπάρχει αυτό. Οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας ήδη προσφέρονται και μάλιστα σε τιμές ανεκτές ε, για τον πολίτη. Έχουμε άμεση κάλυψη. Εάν κοιτάξουμε τις δυνατότητες της LTE, της ε, Fiber to the Home, της ε, παροχής σύνδεσης με νέε ίνε τέλο πάντων στην, στον νοικοκυριό, έχουμε εμεί πολύ ταχύτερη δυνατότητα εξυπηρέτηση. Ε, η διαβάθμιση στις υπηρεσίες και την ταχύτητα εδώ πάλι έχουμε το ψηφιακό μέρισμα με, με την ε, μετάβαση από τη βασική πρόσβαση σε ταχύτητα και την πρόσβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο. Έτσι έχουμε και καλές τιμές και μέχρι και 2 Mbit ε, οπουδήποτε στην Ευρώπη και υψηλής ποιότητας ε, τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και ε, VoIP, Voice over Telephone. Για δε το βίντεο νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη απόδοση της μετάδοσης του περιεχομένου βίντεο από ότι ε, στο δορυφόρο. Εμείς το έχουμε καταφέρει λοιπόν και μπορούμε από τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν τώρα στην αγορά, σε όλη την Ευρώπη, να εξασφαλίσουμε συνδέση ευρυζωνικότητας και συνεχίζουμε με τα 4 Mbit με τις ζώνες που φτάνουν μέχρι τα 10 Mbit και προχωρούμε ακόμη περισσότερο. Ως προς την καινοτομία, ο δορυφόρος αποδείχθηκε πρωτοπόρος πιστεύω και στην ψηφιακή τηλεόραση και στην ψηφιακή μετάβαση. Ο δορυφόρος άρχισε το 96 ήδη με την Canal Sat της Γαλλίας την εφαρμογή αυτή. Και τώρα βλέπουμε ότι το περιεχόμενο στους δορυφόρους είναι κατά 90% πλέον ψηφιακό. Δηλαδή έχει ξεπεράσει κατά πολύ το switchover της επίγειας. Μπορέσαμε επίσης να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου σε υψηλή ευκρίνεια τηλεόραση, χάρη στο δορυφόρο. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο δορυφόρος έχει εξασφαλίσει πολύ σημαντικέ προόδους. Στην Ευρώπη έχουμε 330 οκτώ τέτοιες ε, εφαρμογές συνεχίζεται η εξέλιξη και με την υψηλή ευκρίνεια, τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και με, τους, με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι δορυφόροι για σύνδεση με την Αφρική, την Ασία και άλλα μέρη του κόσμου. Ένα πράγμα που θα πρέπει πιστεύω να υπογραμμίσουμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματο για την αξιοποίηση του φάσματο, θα πρέπει να διατηρήσει το δυναμικό του για ανάπτυξη δυνατοτήτων ή δυναμικού ο Πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται λοιπόν χρόνια για το σχεδιασμό του και την κατασκευή του και έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Έχει περίπου 50 χρόνια διάρκεια ζωής ο δορυφόρος και ω εκ τούτου ε, χρειαζόμαστε ένα σαφές ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε δηλαδή να δούμε κάθε τόσο και αυθαίρετες ε, τροποποίησεις της νομοθεσίας. Δεν θέλουμε ανατροπή του ρυθμιστικού πλαισίου στο οποίο έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Γιατί αυτά που βλέπει ο δορυφόρος ε, το διάστημα δεν περιορίζονται μόνο στην Ευρώπη η συνδεσιμότητα, ιδιαίτερα στο Sinband, με τον υπόλοιπο κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ έχουμε να κάνουμε με υπηρεσίε ευρωπαϊκέ που παρέχουν υπηρεσίε ίντερνετ, επιχειρήσει ευρωπαϊκέ που παρέχουν υπηρεσίε ίντερνετ στην Αφρική. Και θα θέλαμε να παραμείνει διαθέσιμο ένα αρμονισμένο πλαίσιο και η αποτελεσματικότητα στην οποία έχουμε ε, στοχεύσει. Άρα αυτό που ζητούμε είναι να έχουμε ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περιττέρω τι δραστηριότητέ μα για να βοηθήσουμε την Ευρώπη να υλοποιήσει του στόχου τη. Και επίση, για να περιοριστώ στα όσα υπόθηκαν και νωρίτερα, θα αναφερθώ στη ΣΥΣΚΟ και μια μελέτη που δείχνει ότι μεγάλο κομμάτι της ε, ζήτησης για την ευρυζωνικότητα λέτε στο βίντεο και όπως είπατε και εσείς είναι καλύτερη η εκπομπή βίντεο μέσω του δορυφόρου. Χωρί λοιπόν να έχουμε ανταγωνιστική σχέση, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συμπληρωματική μεταξύ των διαφορών τεχνολογιών και ο δορυφόρο μπορεί να προσφέρει το τμήμα του βίντεο στι υπηρεσίε ευρυζωνικότητα. Θα σταματήσω εδώ. Θα ήθελα γρήγορα να επισημάνω ότι υπάρχει μια συζήτηση τροκυλή τραπέζη που οργανώνεται αύριο στο κτίριο εδώ του Κοινοβουλίου από ό,τι γνωρίζω για όποιον ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ πολύ που σεβαστήκατε το χρόνο σας. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Ντενίς Λεσκό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο ίσως το να μιλάει κανείς τελευταίος γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα και ε, ενδιαφέροντα πράγματα. Όταν προετοίμασα την παρουσίαση με τον Ζεράρ Πογκορέλ, τον συνάδελφό μου, επιλέξαμε να δώσουμε μία συμπληρωματική άποψη, συγκεντρώνοντας την προσοχή μας σε κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ και αρκετό καιρό, είναι η ενιαία αγορά των τηλεπικοινωνιών. Συμφωνούμε με πάρα πολλά από αυτά τα οποία ακούσαμε. Συμφωνούμε λέγοντας ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας ε, ε, στη σε κίνηση, νομαδικά σε εισαγωγικά, περνούν τα σύνορα, ταξιδεύουν όλο και περισσότερο και σε ένα τέτοιο θα έλεγα κινητικό πλαίσιο για να επικοινωνήσει κανείς ακόμα και αν υπάρχει Wi-Fi παντού είναι τα κινητά τηλέφωνα που παίζουν ρόλο είτε με το 3G είτε με τα smartphones. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η χρήση της κινητής τηλεφωνίας μπορεί να φανεί σαν ένα στοιχείο το οποίο είναι σε θέση να ενισχύσει την ελευθερία κίνησής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς την δημιουργία μιας ασύρματης ε, με υψηλή ταχύτητα εσωτερικής αγοράς. Ένα βήμα δηλαδή προς τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ενιαίας αγοράς, κάτι το οποίο δεν απασχόλησε πολλούς σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία είναι 27 ακουάριο μέσα στο οποίο κάποια έξυπνα ψάρια όπως ε, είναι και τα έξυπνα τηλέφωνα δεν μπορούν να ξεπερνούν τα σύνορα όπως αυτά θα ήθελαν. Πρέπει να επανέλθουμε σε δυνατότητες επικοινωνίας, πρέπει οι υπηρεσίες να μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα χωρίς προσκόμματα και να διασφαλίζουν μια ρευστότητα της ενημέρωσης για τον καταναλωτή. Το ίδιο σημαντικό και πιο σημαντικό είναι για τον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που ακόμα και αν είναι αναπτυγμένες τοπικά και περιφερειακά θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και ως εκ τούτου έχουν ανάγκη ε, μία πρόσβαση στο σύστημα ενημέρωσής τους, στον κατάλογό τους, στις τράπεζες δεδομένων τους, εν όμως αυτά. Με ικανότητες και με ταχύτητες οι οποίες να είναι ικανοποιητικές, ταχύτητες οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ε, ταυτόχρονη συζήτηση και ενημέρωση και φυσικά με βατό κόστος. Αν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτήν την ενιαία αγορά των τηλεπικοινωνιών και των κινητών, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το φαινόμενο της πολυδιάσπασης της αγοράς που παρατηρούμε σήμερα. Έχω βάλει εδώ κάποιες αποδείξεις θα έλεγα οι οποίες κυκλοφορούν. Βλέπετε μία απόδειξη στη Γαλλία, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. 133.000 ευρώ για ένα μήνα κινητής τηλεφωνίας. Αυτό ήταν πριν από το 2009. Και το 2010 ο William Harrison, ένας Άγγλος, χρησιμοποίησε το κινητό του για broadband στο Παρίσι και βρέθηκε με ένα λογαριασμό 8.000 στερλινών. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πρόβλημα υψηλής τιμολόγησης για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σήμερα παρατηρεί κανείς τρία εμπόδια σε αυτή την ενιαία αγορά και πριν μιλήσω για μια αποτελεσματική διαχείριση του φάσματος. Καταρχάς υπάρχουν επιβαρύνσεις πάρα πολύ ψηλέ όταν ταξιδεύει κανείς από τη μία χώρα στην άλλη και χρησιμοποιεί φυσικά τις δυνατότητες του κινητού του. Αυτό ε, μερικές φορές δημιουργεί πρόβλημα στον καταναλωτή αλλά και στον, ε, στις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να υποστούν αυτά τα κόστη εύκολα και που παρεμποδίζονται μερικές φορές να εργαστούν σε άλλα μέρη στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, και αυτό το είπαν αρκετοί προλαλήσαντες, υπάρχει μια πολύ διάσπαση στο management του φάσματος στην Ευρώπη, υπάρχουν προβλήματα χωρητικότητας, και όλα αυτά αποτελούν επιπλέον προβλήματα. Δεν υπάρχει σαν παράδειγμα μια πανευρωπαϊκή άδεια εκμετάλλευσης που θα επέτρεπε να εξελίσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σχέση με το φάσμα με ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα είναι η δομή των ηλεκτρονικών αγορών μας. Στην ουσία περιλαμβάνει ολιγοπόλια, πάρα πολύ εσωστρεφή, άδειες λειτουργίας και εκμετάλλευσης 15 ετούς ή 20 ετούς διάρκειας, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης που θα διευκόλυνε τις διαδικασίες της καινοτομίας και της ε, αλλαγής σε βάθος της αγοράς. Με άλλα λόγια, ποιες είναι οι αρνητικές πλευρές σε αυτά όλα τα εμπόδια που προέρχονται από όλα αυτά τα εμπόδια. Πρώτον, υποχωρούμε όλο και περισσότερο την δημιουργία αυτή τη ενιαία αγορά των ηλεκτρονικών αγορών. Εγώ εργάζομαι χρόνια στον τομέα αυτό, ακούω για την δημιουργία της ενιαίας αγοράς των τηλεπικοινωνιών εδώ και χρόνια. Το τελευταίο πακέτο τηλεπικοινωνιών το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό, το συζητάμε πολύ, αλλά τίποτα δεν βλέπουμε. Ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά βέβαια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ σημαντικό θέμα, είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στην βάση θα έλεγα της καινοτομίας. Πρωταγωνιστές, μικροί σε μέγεθος, αλλά ευκίνητοι, γρήγοροι, δημιουργικοί, και θα θέσουν αυτά τα οποία έχουν αναπτύξει γρήγορα στην αγορά. Σε αυτή την περίπτωση η πολυδιάσπαση την οποία περιέγραψα προηγουμένως στον τομέα των τιμών και των υπηρεσιών δεν επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο από το σύνολο σύστημα. Ένα παράδειγμα, εγώ δουλεύω σε μια μεγάλη εμπορική σχολή ε, της ε, Γαλλίας και ε, στην ουσία έχουμε ε, κάποιες μορφές συνεργασίας manager με φοιτητέ. Κάποιοι συνεργάζονται στα θέματα της ε, διαχείρισης ε, της ζωής των ηλικιωμένων με ασύρματο τρόπο στο σπίτι τους, στην κατοικία της. Έχουμε λοιπόν μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να να εξάγουν την τεχνολογία τους στην Ευρώπη. Δουλεύουν σωστά στη Γαλλία με την εξαπόσταση διαχείριση των προβλημάτων των ηλικιωμένων, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη δυσκολεύονται να πάνε, ενώ στη ΣΥΠΑ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυκλοφορούν πιο γρήγορα. Ένα άλλο θέμα το οποίο θίγει την κινητικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων κτλ σχετικά με την επαύριο και τις μελλοντικέ δυνατότητες. Πάντα μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα είναι το αύριο. Το αύριο είναι σε 10 χρόνια για μένα. Τι θα γίνεται με τις υπηρεσίες νέας γενεά σε 10 χρόνια. Θα έχουμε συστήματα τα οποία θα υπακούν σαν παράδειγμα που θα επιτρέπουν την χρήση της ενέργειας με πιο αποτελεσματικό τρόπο, θα καλύπτουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες που έχουμε σε σχέση με την αηφόρο ανάπτυξη, με το γραφείο στο σπίτι, με την εκπαίδευση στο σπίτι μερικές φορές κτλ. Έχουμε λοιπόν κάποιες δυνατότητες επέκτασης, έχουμε πιθανότητες εκπαίδευσης, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Εγώ πριν λίγα χρόνια δούλευα στην αρχή εποπτείας των τηλεπικοινωνιών και εκείνη την εποχή κανένας δεν πίστευε ε, ε, τι ακριβώς θα γίνει με το λεγόμενο ψηφιακό ρήγμα. Αν αύριο θέλουμε να υπάρξει ένα παραγωγικό μέλλον με νέες καινοτομίες, με καινούργιες μορφές ε, δράσης, τότε θα πρέπει να είμαστε δεκτικοί ανεξάρτητα της πολιτικής την οποία θα ακολουθήσουμε, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που οδηγούν την καινοτομία. Και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν εργαστήρια, χώροι μελέτης, πειραματικής, έρευνας κτλ. Όλα αυτά λοιπόν πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών που βασίζεται σύμφωνα με εμάς στην ύπαρξη πανευρωπαϊκών ε, ε, επιπέδων χρήσης που θα χρησιμοποιούν τα δίκτυα με ουδέτερο τρόπο έτσι ώστε ο καταναλωτής να μην ψάχνει ε, τον παροχέα της επιχείρησης αλλά να έχει μια ευκολία άμεσης σύνδεσης και χρήσης. Είπαμε, έχουμε την δυνατότητα βέβαια του ψηφιακού μερίσματος ή ψηφιακού κέρδους, το οποίο ε, θα ε, δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, αλλά είναι μια ευκαιρία και για την πρόκληση, θα έλεγα, ε, κατάργησης των ολιγοπολίων, και ταυτόχρονα οι πλατφόρμες αυτές, αυτά τα επίπεδα δράσης μπορούν να ξεκινήσουν την δημιουργία ενός πρώτου σταδίου της ενιαίας τηλεπικοινωνιακής ευρωπαϊκής αγοράς. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με τα πολιτικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, όπως το μέσο της διαχείρισης του φάσματος, και όπως έλεγε ο Φόρτζο λίγο πριν, να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε το φάσμα με δυναμικό τρόπο, έτσι ώστε να γεννήσουμε σε εισαγωγικά νέες υπηρεσίες και να εξαντλήσουμε τις δορυφορικές δυνατότητες όπως έλεγε ο Πίτερ πριν λίγη ώρα. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή σε εκμεταλλευτούμε το φάσμα θα τεθούν δύο ερωτήσεις. Μιλάμε για το ψηφιακό μέρισμα και κέρδος, αλλά δεν μιλάμε για το τι θα συμβεί μετά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν και την ανταγωνιστική ε, διακανονιστική ρύθμιση που θα πρέπει να υπάρξει έτσι ώστε οι τιμές αυτής ε, της δραστηριότητας να μην προσανατολίζονται προς τα πάνω αλλά προς τα κάτω στις οικιακές λεγόμενες τιμές και τα επίπεδα τιμών. Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να ε, ε, εφαρμοστούν θα είναι καταρχάς η τεχνολογική ευελιξία, θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι να κάνουν τις τεχνολογικές επιλογές που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και μια δευτερεύουσα αγορά που θα συνδέει το φάσμα με άλλες τεχνολογίες και με μια κοινή συλλογική χρήση του φάσματος. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης το άνοιγμα της αγοράς, το επαναλαμβάνω. Αν δούμε τι κάνει η Microsoft, η Google, η Amazon, όλες αυτές οι επιχειρήσεις όπως το eBay ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργήσαν σαν, σαν θερμοκοιτίδες θα έλεγα νέων δραστηριοτήτων και να μπορέσουν νέες επιχειρήσεις να μπουν στους χώρους αυτούς και να ε, πολλαπλασιαστούν. Thank you very much. And, um... Σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Αυτά που είπατε για το Google και το Yahoo, ότι εξ αρχής ήταν ε, ε, στην αρχή ήταν μικρές επιχειρήσεις, Ισχύει αυτό. Έχουμε και εμείς στη Σουηδία μια εταιρεία που λέγεται Spotify που θέλει να προσφέρει μουσικές υπηρεσίες, επιπληρωμή. Ριζοσπαστικό θα ακούγεται, έτσι, γιατί κανείς δεν πληρώνει σήμερα, αλλά... Ε, έχουν επιτυχία, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είναι κατακαιρματισμένη η αγορά από πλευρά πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, αντίθετα με τη ΣΥΠΑ. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και τονίσατε όλα αυτά τα προβλήματα. Για να ακούσουμε τώρα, υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Ε, Εγώ θα ήθελα λοιπόν, αφού δεν υπάρχει άλλος εθελοντής, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί παρουσιάζετε τις απόψεις σας, μοιράζεστε τις εμπειρίες της γνώσης σας μαζί μας και κάνατε μια εύκολη σύνοψη. Είπατε ότι είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Δεν ε, ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε το εύρος των αλλαγών. Ε, όλα είναι πολύ περίπλοκα. Ε, ξέρετε, είμαι λίγο ηρωνικός στο ύφος μου. Intervention you listen to or... Αλλά με όλα αυτά τα πάνελ, όλε αυτέ τι ακροάσει μπερδευόμαστε, κινούμεθα σε υψηλά διανοητικά επίπεδα μάλλον, αυτό θα φταίει. λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα πιο από το επίπεδο. Συγκεκριμένα μπορείτε να προτείνετε κάποιες δράσεις, κάποιες αλλαγές για την οδηγία, για ε, περί στην Ολομέλεια. Ξέρετε, εμεί έχουμε δύο λεπτά για να μιλήσουμε κατανότατο όριο. Θα έχετε κι εσεί λοιπόν δύο λεπτά να μα πείτε πώ θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα, προ ποια κατεύθυνση. Κοιτάξτε, ε, το ε, μη αδειοδοτημένο κομμάτι θέλουμε να επεκταθεί στα 5 GHz συγκεκριμένα. Δεν ε, ενοχλεί τους χρήστες και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να το προτείνει αυτό. Πέραν αυτού, επειδή υπάρχει κάτι που δεν συζητήσαμε επί μακρόν και ελπίζω να γίνει στο μέλλον, στο αδειοδοτημένο κομμάτι του φάσματος που είναι εξίσου σημαντικό, θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε τις ε, προθεσμίες όσες έχουν τώρα στο πρόγραμμα της Επιτροπής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε να αρχίσουμε να εξετάζουμε το ενδεχόμενο ε, μελλοντικής περαιτέρω ανακατανομής, αναδιανομής ε, τμήματων του φάσματος. Ο κύριος Χέκμαρκ, μας δείξατε όλες αυτές τις καμπύλες από πλευρά ΣΥΣΚΟ για την αύξηση του όγκου των δεδομένων. Αλλά δεν συζητήσατε καθόλου το θέμα της ταχύτητα, τουλάχιστον όχι σήμερα. Είναι μια άλλη ε, πολύ συζητημένη διάσταση του ζητήματος, ε, γιατί με πέρα από την αύξηση της υπάρχει η αυξανόμενη ζήτηση για ένα και μεγαλύτερη ταχύτητα, πάνω από 100 MB για την περίοδο μετά το 2020. βλέποντα όμω πόσο κατηγιστικέ ήταν οι εξελίξει στο παρελθόν, ε, θα είμαστε ουραγοί. Τι θα έχουμε για το 50% του πληθυσμού το 2020 ταχύτητα 100 MB. Η Νότια Κορέα θα έχει 1000 MB <laughs> για πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της ε, τότε, το 2020. Ε, οπότε απαντήστε μου και εσείς και όλοι, όπως ε, αν λάβετε υπόψη της προτάσεις Επιτροπής και βάση της μεθόδου κατανομής του φάσματος όπως ε, ισχύει σήμερα. Πώς ακριβώς θα ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσει, απάντηση. Ε, η ταχύτητα δεν σχετίζεται μόνο με το φάσμα. Το πρώτο προφανές είναι ότι όσο μεγαλύτερα είναι τα κανάλια μέσα στο φάσμα, ε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ταχύτητα. Όσο περισσότερο φάσμα δώσετε, έτσι, όσο μεγαλύτερη ψαλίδα συχνοτήτων, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα θα έχετε αλλά ε, για την κινητή τηλεφωνία ο στόχος είναι να υπερβούμε ακόμη και τα 40 LT. Αλλά όχι, ε, το 2020 μιλάμε για 100 MB το δευτερόλεπτο, αλλά ήδη απέχουμε πολύ από αυτό. Το σημαντικό πάντως πρέπει να προσθέσουμε είναι οι οπτικές ίνες. But also in the mobile. και για την κινητή τηλεφωνία να την προσαρμόζουμε στην οικιακή χρήση. Δηλαδή, ε, από το, την κεραία μέχρι το σπίτι είναι ασύρματο το δίκτυο. Μετά χρησιμοποιείται το επίγειο δίκτυο. Και αξιοποιώντα αυτό το χαρακτηριστικό μπορούμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη, καλύτερη συγγνώμη, ταχύτητα και καλύτερη χωρητικότητα. Ο κύριος Νίφτρικ. Ευχαριστώ πολύ για να επανέλθω στην ερώτηση. Εμεί δεν ζητάμε να αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Εμείς απλώ ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να λάβουν προσεκτικά υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο και ιδιαίτερα την Ένωση των Διεθνών τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Θα ξέρετε ότι υπάρχει και η KU και η KAKC ζώνες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται. Την ε, KA τώρα, εδώ και πολύ καιρό μάλιστα, χρησιμοποιούν δορυφόροι. Και έτσι προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο τελικό ε, πελάτη. Χάρη στην αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει ο δορυφόρος με την ε, επανάχρηση κάθε 2-3 μοίρες της ολόκληρου του φάσματος, νομίζω μπορούμε να έχουμε τεράστια αποδόση δεν θα σχολιάσω το ζήτημα των 800 MHz γιατί είναι πολύ χαμηλό για μας τόσο όσον αφορά την απόσταση από το διάστημα όσο και ως προς το φάσμα. Αλλά και ναι, μεν το BBC μπορεί να καλύπτει το 90% των πελατών στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το υπόλοιπο 10% που ίσως δεν ε, τα φτάσει ούτε η οπτική ίνα, ούτε άλλου τύπου μετάδοση. Επομένως, η μόνη τους επιλογή παραμένει δορυφόρος. Και αυτή είναι η δική μας δουλειά. Να εξασφαλίσουμε την συνδεσιμότητα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ κύριε Λουσκόπ. Για την πρώτη ερώτηση. όπως είχαμε πει ήδη και στην ε, παρουσίαση, θα πρέπει πιστεύω να θεσπιστούν πανευρωπαϊκές άδειε. Ό,τι τελικά και να γίνει θα μπορούσαμε ασφαλώ να συντονίσουμε το έργο, να συνδυαστούμε και βάση περιπτώσει νομίζω θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ε, ιδέα αυτή της ιστορικής αγοράς. Και τις άδειε, τις λεγόμενες open source που εγώ θα προτιμούσα και εκεί ε, ε, θα έπρεπε να βρεθεί μια διαφορετική λύση για την πληρωμή που καθοδηγεί την αγορά σε ορισμένες επιλογές και την αποστρέφει από κάποιες επιλογές που θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες τις χώρες μας. Επίσης, θα μπορούσαμε να βρούμε ένα σύστημα με άδειες στις ζώνες όπου, για να συμφωνήσω με τον συνάδελφο το SES, e ε, μπορούμε να προσφέρουμε σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές λύσεις να προσεγγίσουμε εμείς τα άτομα αυτά και ναι, μπορεί εκεί ο δορυφόρος να αποδειχθεί πολύ καλό μέσο. Για τη ζώνη των 800 μεγαλύτερα δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Συμμερίζω με τόσο είπαν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και ποιο άλλο θέλει να λέει αυτό, λέω, παρακαλώ. not, um, could... Εάν όχι, ευχαριστώ τα μέλη του πάνελ, του ομιλητέ μα για τη συζήτηση. Έχω, έχω κάποιες σύντομες παρατήρησεις. Ένα από τα πράγματα που προκύπτουν στη συζήτηση είναι ότι χρειάζεται ασφαλώς να εξεταστεί η χρήση των commons, ε, τα, τα χαμηλά σημεία του φάσματος, τα 5 MHz που αναφέρατε εσείς ε, αλλά και άλλοι. Αυτά πρέπει να τα δούμε λοιπόν. Ε, οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες είναι επίσης ένα ενδιαφέρον θέμα. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα πράγματα στο με αυτόν. Αυτή άλλωστε πρέπει να είναι και η βασική πρόθεση της νομοθεσίας που θα προχωρήσει, δηλαδή να καταστεί δυνατή η πρόοδος προς αυτήν την λύση. Δυνατότητες και άδειες κοινέ. Και περνάμε στη συζήτηση για το πώς μπορεί να ανοίξει αρκετό μερίδιο του φάσματος. Υπάρχει πιστεύω μια τάση και αυτό σαν απάντηση στην συνεχιζόμενη συζήτηση, στην εξελίξη συζήτηση. Διότι βέβαια δεν έχω καταλήξει την έκθεσή μου, θα την υποβάλω στην... Ε, ε, Επιτροπή το, στα τέλη Φεβρουαρίου. Άρα δεν έχω κατασταλάξει. Αλλά θέλω να πω το εξή, ότι εάν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί είναι γνωστό ότι η Ευρώπη χρειάζεται 1200 MHz συνολικά. Και τώρα έχουμε φτάσει στα 800 νομίζω. Μάλλον είμαστε στη ζώνη των 800, έχουμε φτάσει στα 500. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε όταν έχουμε όχι μόνο αύξηση στις, ε, στην ε, ε, κυκλοφορία αλλά και στις υπηρεσίες. Είδα Φερρυπίν πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει τις εξελίξεις. Βλέπουμε καθημερινά σχεδόν ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα όρια της τεχνολογίας, ούτε το iPhone, ούτε το iPad έχουν πει τελευταία λέξη. Κάθε βήμα θα φέρει ένα καινούριο και μια νέα πρόοδο. Άρα... Θα χρειαστεί μάλλον να έχουμε μια ανοιχτή προσέγγιση. γιατί ασφαλώς δεν γνωρίζουμε τι θα προκύψει. Μερικέ φορέ θυμάμαι την εποχή που είχαμε την ασπρόμαυρη τηλεόραση και λέγαμε τι υπέροχο πράγμα αυτή η τηλεόραση. Και όντω ήταν υπέροχη. Αλλά δεν ξεπέρασε τεχνολογία. Όλοι νομίζω συμφωνούμε και θα συμφωνήσουμε Πασίλτος πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις εξελίξεις. Και στο τελευταίο να έχουμε μια ματιά και προς τις αλλαγές του 80 και το 90 και το ε, κινητό τηλέφωνο που εμφανίστηκε τότε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους όσοι λάβατε μέρος σε αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.